So, liebe Kollegen, Kollegen, können wir beginnen? Αρχίσουμε, συνάδελφοι. Wir haben den Punkt 16 aufzurufen. Έχουμε το σημείο 16. Ακαιρεότητα και διαφάνεια της ενεργειακής αγοράς. Η αρμόδιος για την έκθεση αυτή που θα τη δούμε έτσι λίγο στα γρήγορα είναι ο συνάδελφος ο κύριος Χατζημαρκάκης που είναι εδώ και ε, να του δώσω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για το REMIT, τον κανονισμό δηλαδή για την ε, διαφάνεια και κεραιότητα της αγοράς ε, ενέργειας ε, που λένε στα αγγλικά και μιλάμε για ενεργειακά προϊόντα που σχετίζονται με το εμπόριο της ενέργειας τα οποία πρέπει να τα δούμε ξεχωριστά γιατί ξέρουμε όλοι πως είναι απαραίτητο να βλέπουμε τις χρηματαγορές διαφορετικά από ό,τι στο, στο παρελθόν ξέρετε πως ε, το 2003 είχαμε την οδηγία περί κατάχρησης δεσπόσας θέσης, οπότε πάντα υπήρχε κάποια ρύθμιση, αλλά ήδη από τότε υπήρχε εξαίρεση για τον τομέα της ενέργειας. Και θέλουμε να τη διατηρήσουμε. Δεν είναι απλό αυτό, γιατί ο Επίτροπος Έτιγκερ που θα έρθει αργότερα συμφωνεί με όλο τον κλάδο πως ε, μία εξαίρεση, ο Remit, χρησιμοποιείται ως ε, λέξη specialis. Υπάρχει η... Υπάρχουν σχετικές οδηγίες, υπάρχει η MIFID, υπάρχουν πάρα πολλοί γάμισμε. Και δυστυχώς υπάρχει δυνατότητα να εκμεταλλευτεί κάποιος τα παραθυράκια. Εξού και ε, το ρέμι το οποίο παρουσιάζουμε. Γιατί τώρα συγκεκριμένα για την ενέργεια. Γιατί πάρα πολύ παίκτες στην αγορά όταν ασχολούνται με παράγωγα της ε, ενέργειας ε, δρούν πάρα πολύ Ε, ανεξέλεγκτα. Δηλαδή, αν το κάναμε αυτό με τις ίδιες απαιτήσει που κάνουμε για τις... αν τους μεταχειριζόμασταν όπως μεταχειριζόμασταν τι τράπεζε, θα έπρεπε να έχουν ε, ε, ίδιο κεφάλαιο, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει, και επιπλέον ο όγκος αυτών των συναλλαγών σχετίζεται με απτά προϊόντα, δηλαδή το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα και Ποιο είναι τώρα ο τομέας. Εδώ πέρα να επικεντρωθούμε, εμεί λέμε, στις ε, αγορές ρεύματο και φυσικού αερίου γιατί έχουν ευρωπαϊκή διάσταση και διαβουλευτήκαμε για το εάν θα έπρεπε να δούμε και το πετρέλαιο και τον άνθρακα αλλά καταλήξαμε στο ότι εκεί πέρα είναι παγκόσμιες οι εμπορικές ροές οπότε μπορούμε να τα παρατηρούμε αυτά τα δύο αλλά όχι να καλυφθούν εδώ πέρα. Διαφορετική είναι η κατάσταση με το διοξείδιο του άνθρακα, δηλαδή το ETS, γιατί έχει μικρή σχέση με το ρεύμα και το φυσικό αέριο και μετά από συζητήσει με την Κομισιόν που έχει τρεις γενικές διευθύνσεις και ασχολούνται με αυτό το θέμα, αγοράς δηλαδή ενέργειας και κλίματος, να βρουν μια λύση. Και θα παραμείνει δηλαδή αυτό το θέμα αρμοδιότητας του ETS και θα υπάρξει μια παρατήρηση η ΕΣΑ η οποία είναι μια υπηρεσία που έχει δημιουργηθεί με το τρίτο πακέτο ενέργειας η οποία θα δει το εμπόριο διοξίδιου του άνθρακα Το πώς ακριβώς θα το δούμε. Τι θα γίνει λοιπόν τώρα με την ΕΣΑ. Η ΕΣΑ είναι μια υπηρεσία Η ΕΣΑ λοιπόν είναι μια υπηρεσία η οποία στο μέλλον θα ερευνά συναλλαγές ε, και θα λαμβάνει ειδοποίηση για όλες τις ε, συναλλαγές ε, φυσικού αερίου και ρευματο και αυτό θα γίνεται είτε μέσω των χρηματιστηρίων είτε από τους εναλλασσομένους όταν είναι εκτός των χρηματιστηρίων, over the counter που λέμε. Και βεβαίως ε, αυτό μπορεί να γίνει ε, όπως γίνεται παραδείγματος χάρη στη Γερμανία όπως στην υπηρεσία ε, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού έχουμε ένα ειδικό παρατηρητήριο της ενέργειας και γίνεται η πρόταση η υπηρεσία αυτή να συλλέγει τα στοιχεία στην θέση της Acer και να τα διαβιβάζει στη Λιουμπλιάνα έτσι ώστε οι συμμετέχοντες στην αγορά τους οποίους ορίσαμε κάπως καλύτερα γιατί ο ορισμός ήταν το 2003 να μην ε, στέλνουν ε, δύο φορές τα ίδια στοιχεία. Όταν λοιπόν ε, λάβει αυτά τα στοιχεία η Acer θα πρέπει βεβαίω να καταλάβει πως είναι ειδικού χειρισμού, είναι κάπως ευαίσθητα, υπάρχουν απαιτήσει εμπιστευτικότητας και από νομική σκοπιά και τεχνική γιατί τα ζητήματα του software ακόμα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Επίσης όταν μιλάμε για δημοσίευση αυτών των δεδομένων θα μπορούν να δοθούν μόνο σε συγκεντρωτική μορφή. Ελπίζω να συμφωνούμε εδώ πέρα με την Κομισιόν. Ποιος καλύπτεται λοιπόν εδώ πέρα. Ο κάθε συμμετέχον στην αγορά ακόμα και όταν ε, δεν έχει μεγάλο ποσοστό θα καλύπτεται. Χρειάζεται λοιπόν ένας κανονισμός για τα επιέλατον όπως λέμε, τα de minimis, και το όρισε η ομάδα ε, εργασίας του Συμβουλίου στα 600 γιγαβατόρες αλλά δεν θέλουμε να το ορίσουμε ως ε, κατόφλι γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς ε, ακόμα. Οπότε θα μπορούσε να γίνει με μια πράξη εξουσιοδότηση και να αφήσουμε μετά στην Κομισιόν να ορίσει ε, το όριο κατά το οποίο θα ισχύουν οι διατάξεις του επιέλατων. Θα δούμε λοιπόν πώς θα τα αντιμετωπίσει αυτά το Συμβούλιο και εμείς. Υπάρχει όμως ένα μνημόνιο μεταξύ μας μνημονιοσύνη αντίληψης μεταξύ ε, των θεσμικών οργάνων για το τι θα γίνει με τις πράξεις ε, κατά εξουσιοδότηση και θα προσπαθήσουμε με την διοργανική αυτή συμφωνία που έχουμε να κάνουμε κάποιο καλύτερο τον ορισμό για τις ε, πράξεις κατεξιότητας και αυτό θα το δείτε και στις τροπολογίες. Τώρα τι γίνεται όταν οι συμμετέχοντες στην αγορά που είναι πάνω από το όριο αυτό, de minimis, στέλνουν τα δεδομένα στη Λιουμπιάνα ή στην Εθνική Υπηρεσία. Και τι γίνεται αν υπάρχει υποψία περί συνεννόησης ε, ε, η κατάχρησης ε, της αγοράς ή εσωτερικής πληροφόρησης. Σε αυτή την περίπτωση η Acer ε, ειδοποιεί τις εθνικές αρχές, οπότε είναι σαφές πως πρέπει πρώτα να κινητοποιηθούν οι εθνικές αρχές, γιατί γνωρίζουμε πως σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και τους διαφορετικούς εθνικούς κανόνες, δεν έχει, αν θέλετε, και τις απαραίτητες αρμοδιότητες ε, για να επιβάλλει κυρώσει κάθε υπηρεσία. Δηλαδή, στη χώρα την οποία γνωρίζω βεβαίως, η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι αρμόδια, αλλά το αποφασιστικό είναι να οδηγηθούμε σε μια εναρμόνιση των κυρώσεων, γιατί πρέπει να αποφύγουμε το εξής. Το να υπάρχει διαφορετικό επίπεδο ποινών και να πάει άρα το εμπόριο εκεί όπου δεν υπάρχουν ποινές ή είναι χαμηλότερες. Οπότε χρειάζεται να έχουμε ενιαίες ε, κυρώσεις. Ανέφερα ήδη τους ορισμούς, ε, οι ορισμοί επικαιροποιούνται και Πρέπει να πω πως η πρόταση της Κομισιόν ήταν ήδη σε πολύ καλό επίπεδο, ήταν πάρα πολύ καλή. Οπότε το θέμα είναι λίγο να τα προσαρμόσουμε χρονικά. Ένα θέμα το οποίο ετέθη και δεν υπήρχε στην πρόταση ήταν η αδειοδότηση. Κάθε συμμετέχον ε, της αγοράς πρέπει να λαμβάνει άδεια ή όπως είπαμε ήδη με τους σκιώδεις ηγητές, πρέπει μόνο να καταγραφεί. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Στο Συμβούλιο υπάρχουν ομάδες που δεν προβλέπουν ούτε καν καταγραφή. Εμείς λέμε τουλάχιστον μια καταγραφή σε εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα θέλαμε. Και όπως σας είπα, καταγραφεί μόνο αν περνάνε το κατόφλι αυτό του de minimis. Και το θέμα είναι τι γίνεται με τα μέρη εκείνα που υπάρχει εμπόριο και είναι σημαντικά ε, σημαντική κόμβη εμπόριο, δηλαδή Νορβηγία, Ελβετία. Η Νορβηγία καλύπτεται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο Η Ελβετία όμως όχι. Οπότε είμαστε ακόμα σε διαπραγματεύσεις και ζητήσαμε από την Κομισιόν για να συμπεριληφθεί και η Ελβετία γιατί περνάνε σημαντικές ροές ενεργειακών παραγόγων από εκεί. Κάτι τεχνικό εδώ πέρα. Είπαμε στον ορισμό πώς θα χρησιμοποιήσουμε παραδείγματα, γενικά παραδείγματα για να εξηγήσουμε π.χ. τι είναι εσωτερική πληροφόρηση από πλευράς, ε, από πλευράς νομοθέτη, για να μην αφήσουμε πολύ περιθώριο ερμηνείας. Οπότε νομίζω πως έτσι όσο έχει το κείμενο είναι καλά και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις ε, συγητές και ειδικά τον κύριο Γκέμπελς ο οποίος έγραψε γνωμοδότηση για την Επιτροπή Οικονομικών η οποία θα είχε λόγους να απορρίψει το Lex Specialis ο κύριος Μπαρινιέ δεν έχει πιστεί ακόμα ότι χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο αλλά εμείς στο Κοινοβούλιο θεωρούμε πως και η Επιτροπή Οικονομικών θεωρεί πως χρειαζόμαστε μια τομεακή προσέγγιση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Να δώσω τον λόγο στον κύριο Γκέρκ, τον Συγητή. Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν ε, να συγχαρώ τον εισηγητή μας ε, για την εξαίρετη εργασία του και τον ευχαριστώ επίσης ε, για την προσπάθεια που κατέβαλε προκειμένου να συνεργαστεί με τους σιώδης ηγητές ευθύς εξ αρχής της όλης διαδικασίας. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ε, έκθεσή του, πρέπει να ομολογήσω πως ε, και εγώ συμφωνώ με την ε, αρχική πρόταση της Κομισιόν. Εμείς τώρα τονίζουμε κάποιους τομείς που θεωρούμε πως είναι και οι σημαντικότεροι. θα τα αναφέρω αυτά εντάχει. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ πως χρειάζεται ένα, ένας λέξ πετσάλης και επίσης ε, συμφωνώ πως ε, χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν οι πράξεις κατεξιοδότηση και αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η, τώρα, η χρηστή διαχείριση των ε, δεδομένων είναι κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνο πρέπει να αποφύγουμε την παράλληλη ε, υποβολή των δεδομένων προκειμένου να υπάρξει μια αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στα κρατημέλη. Αυτά λοιπόν είναι τα σημεία που θα ήθελα να θίξω και να δηλώσω ότι συμφωνώ επί όλων αυτών των σημείων όπως αυτά αναφέρονται στην έκθεση. Τώρα έχω πέντε ζητήματα που με απασχολούν και θα ήθελα εντάχει να τα αναφέρω. Πρώτα απ' όλα ε, ό,τι αφορά την ε, διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή ε, τη οδηγία. Μιλήσαμε για το, πετρό, πετρέλαιο και τα παράγωγα και για το διοξείδιο του άνθρακα. Και για τα δύο ζητήματα πραγματικά ανησυχώ. Δεν μπορώ να φανταστώ την διεύρυνση προς το πετρέλαιο και τα παραγωγά του. Πρόκειται για αγορές πολύ διαφοροποιημένες. Υπάρχουν συγκεκριμένες για αυτά τα ζητήματα και υπάρχουν παράμετροι εντελώς διαφορετικοί που ισχύουν για τον ηλεκτρισμό και για το αέριο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να υπάρξει ενημέρωση πάνω στο ζήτημα. Τώρα, ε, το ζήτημα της ε, εμπορίας εκπομπών ε, το κατανοώ αλλά θεωρώ ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Τώρα, η ανταλλαγή εκπομπών ε, είναι πιθανό να οδηγήσει σε κάποιες καταχρήσεις διαφορετικές από αυτές που αφορούν ε, τις απάντες στον τομέα του ηλεκτρικού ρεύματος, ε, του αερίου κλπ. που άπτονται περισσότερο θεμάτων ΦΠΑ. Προς το παρόν δεν έχει εξευρεθεί κάποια απάντηση σε αυτό το πρόβλημα των καταχρήσεων. Εξάλλου, δεν ε, θα ήταν εύκολο να καλύψουμε όλο το πεδίο που θα αφορά τις ανταλλαγές εκπομπών. Χρειάζεται να παρακολουθούμε κάποιους τομείς όπως τον τομέα της βιομηχανίας της Ζαχάρεως ή της Ιάλου. Είναι πολύ περίπλοκο να το πετύχουμε και ως εκ τούτου θα είναι δύσκολο να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά το σύστημα όπως αρχικά πιστεύαμε πως θα μπορούσε να συμβεί. Αν θέλουμε λοιπόν να ρυθμίσουμε και το θέμα των ανταλλαγών εκπομπών υπάρχει ανάγκη από μια οδηγία ad hoc. Χρειάζονται διάφοροι μηχανισμοί, χρειάζονται μελέτες αντικτύπου κλπ. Κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνο, αλλά να το εισαγάγουμε έτσι χωρίς προηγούμενη προετοιμασία νομίζω ότι είναι κάτι αμφιβόλου αποτελέσματος. Τώρα κάτι άλλο που με απασχολεί, το θέμα των ε, αδειοδοτήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ως στόχο με βρίσκει σύμφωνο. Άδειε οι οποίε θα είναι ισότιμε και θα σχήμα το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δημιουργία μια ε, κοινή ε, αγορά ηλεκτρισμού. Αλλά το ζήτημα αυτό το μα ταλανίζει εδώ και μια δεκαετία και δεν έχουμε κατορθώσει να ξέρουμε τι Λοιπόν, εάν αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας, ε, αυτού του κανονισμού, είναι πιθανόν ε, να διακυβευτούν οι αρχικοί στόχοι του κανονισμού. Χρειάζεται να βρούμε μια χρυσή τομή. Συμφωνώ με τον εισηγητή που αναφέρθηκε στον, ε, στην καταγραφή, αυτό το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει έναν συμβιβασμό, δηλαδή να αντικαταστήσουμε την άδεια με την καταχώρηση και ένα τρίτο σημείο που μου δημιουργεί αμφιβολίες είναι αυτό της εναρμόνισης των κυρώσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μια ακόμα φορά θα να πω ότι ως στόχο με βρίσκει σύμφωνο η πρόταση. Δηλαδή, ε, στη θεωρία μπορώ να τον στηρίξω, αλλά Εάν δεν κατορθώσουμε να επιτύχουμε το στόχο, τότε ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός, όπως πολύ ορθά είπε και ο εισηγητής. Δεν γνωρίζω όντω ποιε είναι οι πιθανότητες να καταλήξουμε σε μια τέτοια εναρμόνιση στο πλαίσιο του Συμβουλίου, διότι με αυτόν τον τρόπο ε, μπλεκόμαστε, θα έλεγα, στα πόδια των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και εδώ διαβλέπω το κίνδυνο αν επιμείνουμε ιδιαίτερα πάνω στο σημείο αυτό να διακυβεύσουμε το σύνολο της εκθέσεως. Γι' αυτό λοιπόν ήθελα να θίξω αυτά τα ζητήματα. Τώρα, ε, συμπερασματικά, για τα δύο σημεία που δεν έθιξε ο συγκητής, αλλά θα ήθελα να αναφέρω πρώτα απ' όλα σε ό,τι φορά τα γραφεία αντιπροσώπευσης. Ε, και εδώ έχω κάποιες αμφιβολίες. Γνωρίζω ότι η υπηρεσία της Λουμπλιάνα συστάθηκε και ξεκίνησε ήδη να, ε, ε, να δουλεύει και τώρα μιλάμε για τη σύσταση νέων ε, γραφείων. Αυτό θα αυξήσει την γραφειοκρατία και αυτό ενέχει κάποιους κινδύνους. Πρέπει να σκεφτούμε αν είναι απαραίτητο να ιδρυθούν αυτά τα νέα γραφεία, αυτές οι νέες υπηρεσίες ειδικά ε, ότι οι πληροφορίες μπορεί να ανταλλάσσονται με ηλεκτρονικό τρόπο, τρόπο μέσω διαδικτύου κλπ. Τα νέα γραφεία, νέε υπηρεσίε χρειάζονται νέου υπαλλήλου, νέα στελέχωση, περισσότερη γραφειοκρατία κλπ. Πρέπει να έχουμε κατά νου τον αρμόδια υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών που για μας μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, ε, υπάρχουν ε, παρόμοιες ε, οργανώσεις και ίσως θα πρέπει να εμπνευστούμε από τη λειτουργία τους. Και τέλος, το ζήτημα των trade repositories. Θα πρέπει να υπάρξουν αυτές οι υπηρεσίες πέραν των υπηρεσιών που ήδη παρέχονται και το, η ρυθμιστική αρχή θα ε, διαδραματίζει ταυτόχρονα και έναν εμπορικό ρόλο. Αλλά αυτό είναι κάπως παρακινδυνευμένο κατά τη γνώμη μου. Αλλά και δεν είμαι σίγουρος αν θα χρειαστεί να αναλάβουμε αυτόν τον κίνδυνο. Αυτές είναι λοιπόν οι ανησυχίες μου, αλλά γενικά θέλω να πω ότι η έκθεση είναι εξαιρετική και πιστεύω πως στο ε, πλαίσιο της πρώτης ανάγνωσης ε, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε για αυτό προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των αγορών. Wir haben ganze Wälder vernichtet, um, um die ganzen Dokumente heute auszudrucken. Ένα δάσος κόψαμε για να τυπώσουμε τα έγγραφα. Μα εσύ τα τύπωσες μόνος σου, λέει ο πρόεδρος. Εσύ, εσύ το κόψεις το δάσος. Αιώνιος αμαρτωλός ενώπιον των δέντρων. Συγχαρητήρια, εν περιπτώσει. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό τομέα, την αγορά ρεύματος ε, και αερίου και ενέργειας και δύσκολο για τους πολιτικούς. Γιατί ποιος από μας ξέρει τι γίνεται στα χρηματιστήρια. Κανείς δεν ε, έχει βρεθεί σε μια συναλλαγή over the counter. Είναι δύσκολο είτε μιλάμε για την υπάρχουσα νομοθεσία είτε για μελλοντική νομοθεσία όπου μιλάμε και για μύφιντ και τα λοιπά. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ποιος μας ψιθυρίζει και μας λέει πραγματάκια στροπολογίες. Να πω λοιπόν κάποια πράγματα. Αυτό το οποίο δεν μου αρέσει απέναντι από την πρόταση της Κομισιόν η οποία φροντίζει να πάνε απευθείας τα δεδομένα στην Acer διακινδυνεύουμε αν αρχίσουμε να λέμε α, να το στείλουμε στη Γερμανία στην υπηρεσία τάδε ή οι οικονομικές πληροφορίες να πάνε πρώτα στις οικονομικές αρχές και μετά στην Acer θα γίνει μετά ένα ψηφιδωτό. Γιατί πώς μπόρεσαν να ανακαλύψουν οι Αμερικάνοι τα εγκλήματα στην αγορά του αερίου. Γιατί σε μια πρόταση κάλυπταν και τις πραγματικές ροές και τις αγορές spot και τις λοιπές ε, αγορές. Και πρέπει να έχουμε λοιπόν μία υπηρεσία, να έχει μία γενική εικόνα, η Acer, όλες οι πληροφορίες πρέπει να γίνουν απευθεία εκεί και εκεί πέρα να γίνεται η κατανομή. Βεβαίω, λένε κάποιοι τεράστια γραφειοκρατία κτλ. κτλ. Πρέπει να ξέρουμε όμως πως υπάρχει ένα πιλωτικό έργο της e-control με τα χρηματιστήρια του Λονδίνου και Φραγκφούρτης και αλλού και εκεί πέρα ξεκαθαρίστηκε πως 90% των πληροφοριών είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Οπότε η παραπάνω προσπάθεια για να πάνε απευθεία στην Acer ταυτόχρονα, δηλαδή στην εποχή του υπολογιστή δεν, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Οπότε προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να πάμε. Σημαντικό είναι να ρίξουμε φως στις συμφωνίες over the counter που δεν καλύπτονται σήμερα. Είναι μικρότερο ποσοστό ίσως ως αριθμός, αλλά αποτελούν το μεγαλύτερο κίνδυνο. την ε, τροπολογία 17 και τον τελικό χρήστη. Και εμείς θεωρούμε πως κάποιοι μεγάλοι τελικοί χρήστες πρέπει να καλύπτονται λόγω του όγκου κατανάλωσης. Οπότε χαιρετίζουμε εδώ πέρα την τροπολογία αυτή και πράγματι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι συναλλαγές over the counter. Για τις άδειε. Πρέπει να ομολογήσω πως είμαι κάπως διχασμένος, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Αν κάνουμε εθνικές άδειε, αυτό σημαίνει πως κάθε ένας που έχει εθνική άδειο πάει στην ε, ευρωπαϊκή ε, αγορά. Άρα τι έχουμε, ελάχιστες προδιαγραφές ή να δώσει τις άδειες η Acer και στις σχετικές τροπολογίες υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που πάνε πάρα πολύ κοντά στις απαιτήσει του ΕΦΕΤ και των ε, εμπόρων και δεν ξέρω πως ανοίγουμε θύρες οι οποίες καλό θα ήταν να Κατόπιν αυτή η ισορροπία μεταξύ Ρέμετ και Ματ και Μίφιντ των οδηγιών των διαφόρων. Στις ε, συζητήσεις που είχαμε έχουμε την αίσθηση πως υπάρχει η τάση να πούμε πως θα κάνουμε τη Remit τόσο μεγάλη ώστε οι μεγάλες εταιρείες αερίου και ρεύματος δεν θα εμπίπτουν στη MIFID. Εμεί θεωρούμε πω για του μεγάλους εμπόρους και τις μεγάλες εταιρείε χρειαζόμαστε και τα δύο. Γιατί ε, είναι τέτοιου μεγέθους ώστε πρέπει να τις παρακολουθούν και οι οικονομικές αρχές και χρειαζόμαστε και όλες τις πληροφορίες για να εμποδίσουμε παιχνίδια στην αγορά. Δεν πρέπει δηλαδή να τους δώσουμε το πρόσχημα να μας πούν πως ε, κοιτάξτε εμείς δεν εμπίπτουμε στη MIFID, είμαστε στη REBIT. Γι' αυτό πρέπει να συνοηθούμε με τον Ρόμπερτ Γκέμπελς και να δούμε με την εμπειρία του τι θα, πώς θα το κλείσουμε αυτό το θέμα. τώρα οι αρχές θεωρώ πως είναι ξεκάθαρη η Κομισιόν και όσον αφορά τη γερμανική ιδιαιτερότητα δεν πρέπει να τη βάλουμε στις τροπολογίες μας. Δεν έχει κανένα νόημα, μόνο προβλήματα δημιουργεί. Εάν κάποια στιγμή στο τέλος των διαπραγματεύσεων ε, χρειάζεται εξαίρεση για τη Γερμανία ή λέξη specialis να το κάνουμε, αλλά να μπει στην έκθεσή σου και στη διαπραγματευτική θέση του Κοινοβουλίου δεν το βρίσκω σωστό. Ε, πρέπει να μείνουμε στην πρόταση Κομισιόν. Η Acer πρέπει να έχει ισχυρό ρόλο. Εγώ θεωρώ πως το Συμβούλιο προσπαθεί εδώ πέρα να μην το κάνει αυτό. Πρέπει λοιπόν να επικρατήσουμε εναρμόνιση των ποινών επίσης πάρα πολύ σημαντική και μπορούμε να αναφέρουμε εδώ πέρα το παράδειγμα της οδηγίας roaming. Επίσης τελευταία δύο πράγματα περιφερειακές αγορές υποθέτω πως για τα επόμενα χρόνια θα έχουμε περιφερειακές αγορές και άρα οι περιφερειακές ρυθμιστικές αρχές είναι πάρα πολύ σημαντικές και αυτό το οποίο δεν βλέπω εγώ είναι πως έχουμε την Acer και τις εθνικές αρχές πιθανώς η συνεργασία ρυθμιστικών αρχών Γερμανίας Γαλλίας και Μπενελούξ και της ε, πενταμερούς αγοράς κτλ. θα αποτελέσει κάτι το σημαντικό. Και πρέπει να σκεφτούμε μήπως ε, θα μπορέσουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στο περιφερειακό επίπεδο γιατί αυτή θα είναι η πραγματικότητα της αγοράς. Τέλος για το διοξείδιο του άνθρακα. Αντιλαμβάνομαι τις αντιρρήσεις του κύριου Γιέργα, αλλά από την άλλη το διοξίδιο του άνθρακα είναι συστατικό του εμπορίου του ρεύματος και πρέπει να φροντίσουμε η Acer να έχει όλα τα δεδομένα γιατί εκεί πέρα προσφέρεται και θα είναι πολύ απλή υπόθεση τα μαγειρέματα. Ούτως ή άλλως στην πρώτη ανάγνωση είμαστε. Ε, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω στη διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ. Σιμάνσκι. Ευχαριστώ To jest oczywiście bardzo poważne sprawozdanie, ponieważ... Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό το έγγραφο που έχουμε αναχείρας και υπάρχει ήδη όμως ε, έγραφο, ε, υπάρχουν έγγραφα ήδη που ρυθμίζουν αυτό το ζήτημα σε διαφορετικούς κλάδους. Πρώτα απ' όλα, να πούμε κάτι σχετικά με την προστασία της εμπιστευτικής προφορίας και πώς δημοσιεύονται αυτές οι εμπιστευτικές προφορίες. Πρέπει να το εξετάσουμε, διότι αφού διάβασα το έγγραφο της Κομισιόν, δεν κατάλαβα απόλυτα τι ακριβώς θα κάνουμε με τους διάφορους ορισμούς, διότι οι πληροφορίε αυτέ ε, δεν αντιμετωπίζονται με έναν και ενίο τρόπο. Αυτέ οι πληροφορίε είναι ευαίσθητε, είναι ε, από εμπορική σκοπιά και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν θα τι χειριστούμε. Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικές οι προτάσεις που γίνονται αναφορικά με τους ε, κανόνες ε, που αφορούν στις πληροφορίες. Ε, οι κανόνες επιθυμούν να ενισχύσουν περαιτέρω το ισχύον σύστημα. Επίσης, ε, είναι, εδώ εμπλέκεται και το ζήτημα της ευθύνης, αλλά και το θεσμικά ζητήματα. Κατά την άποψή μου, το πρωτόκολλο συμφωνίας που αφορά στις ε, κατεξοδότηση πράξεις είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να μας καθοδηγεί. Θα πρέπει στο, να δούμε στο μέλλον πώς δεν θα έχουμε προβλήματα όταν η Κομισιόν θα περάσει στην εκτέλεση αυτών των ε, κατεξοδότηση πράξεων. Όλες αυτές οι προτάσεις ε, τείνουν στο να βελτιώσουν η κατάσταση δίνοντα περισσότερε αρμοδιότητε στο Κοινοβούλιο. Αλλά εμεί πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τώρα σε ό,τι φορά τι ε, κυρώσει και τι ε, διαδικασίε. Ε, τα όσα αναφέρονται εδώ είναι σωστά. Αλλά δεν θα θέλαμε να έχουμε μια πολύ καλή νομοθεσία η οποία όμως δεν θα μπορεί στην ουσία να εφαρμοστεί. Πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες ε, των εθνικών Διεθνιστικών αρχών ενέργειας. Ταυτόχρονα πρέπει να μας αποσχολήσει το ζήτημα της εφαρμογής των κυρώσεων. Πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο αναφορικά με τη διαδικασία που θα ακολουθεί. Και κάτι ακόμα. Εδώ εξετάζεται η όλη δομή της ε, υπηρεσίας ΑΣΕΡ ε, αναφορικά με την ε, οργάνωση, με τα περιφερειακά γραφεία, περιφερειακές υπηρεσίες ε, και όλα τα μέσα τα οποία παρέχονται. Αυτά τα μέσα πρέπει να παρέχονται στην κεντρική υπηρεσία. Δεν θα πρέπει τώρα να αρχίσουμε να κατακαιρματίζουμε αυτά τα μέσα και αυτά τα κονδύλια τα οποία έχουμε και χορηγούμε στην ΑΣΕΡ. Τώρα σε ό,τι το REMIT ε, θα πρέπει να προσέξουμε το θέμα της ε, εμπορίας ε, εκπομπών και της ανταλλαγής εκπομπών αλλά υπάρχει και κίνδυνος να διευρύνουμε περαιτέρω την όλη νομοθετική διαδικασία κάτι το οποίο θα δυσκολέψει την εφαρμογή των ε, κανονισμών. Να η έκθεση μας βρίσκει σύμφωνος. Ε, το Ρέμιλ θα μπορούσε να περάσει στο πλαίσιο της πρώτης ανάγνωσης ε, και ελπίζουμε πως με τη συνεργασία των εισηγητών και των σχεδόν εισηγητών το θέμα θα προχωρήσει άμεσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τον εισηγητή, τον κύριο Χατζή Μαρκάκη, διότι έχει βελτιώσει σημαντικά το αρχικό κείμενο της Κομισιόν και επιθυμώ να αναφερθώ σε κάποιες ιδέες της εκθέσεως Τώρα, πέραν των ανησυχιών σε ζήτημα ασφάλειας δικαίου, θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση σαφή σχετικά με ποιες θα είναι οι πράξεις οι οποίες θα δημοσιεύονται. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω στο σκεπτικό 5, 9 των άρθρων 5 και 8 θα ήθελα να καταστήσω σαφές ή συγκεκριμένος τύπος ε, δημοσίευσης θέτει τέρμα στην ε, inside information, στις ε, πληροφορίες που κυκλοφορούν στο εσωτερικό, όπως, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5.1. Θα ήταν παρακεντρευμένο να θεωρήσουμε ότι η πληροφορία είναι δημόσια, είναι κοινή, όταν δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο με θέματα που αφορούν το trading, την εμπορία και τα μέσα ενημέρωσης. Επίσης, έχω εμβολίες αναφορικά με το θέμα της ασφάλειας δικαίου και τον συνδυασμό με την έννοια της προσπάθειας χειραγώγησης όπως αναφέρεται στο δεύτερο άρθρο, παράγραφοι 2 και 3 και στο άρθρο 3, παράγραφος 4 πώς ε, μπορούμε να αποδείξουμε την προσπάθεια χειραγώγησης. Είναι κάτι που από νομική σκοπιάς ε, είναι ασαφές και πρέπει να το διευκρινίσουμε περαιτέρω. Τρίτον, να τονίσω πως ε, οι τιμές της αγοράς δημιουργούνται από την ε, ζήτηση και την προσφορά και άρα επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες. Το χρόνο, τις συνθήκες συντρολογικές, ε, τον ε, ανέμους, το δίκτυο διανομής, μεταφοράς κλπ. Οι επιπτώσεις της ζήτησης επί των τιμών ε, είναι κάτι που χρειάζεται να αναγνωριστεί πλήρως στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής ως ε, μία από τις βασικές αιτίες ε, του καθορισμού των τιμών. Και τώρα στο αναφορά στο κόστος, το καθαρό κόστος μεταφοράς στο σκεπτικό 10, το λογική σκέψη 10, νομίζω ότι είναι ανεπαρκές διότι δεν λαμβάνει υπόψη το διάφορες ε, δαπάνες ε, με που είναι απαραίτητες μέχρι να ξεκινήσει να λειτουργεί ένα εργοστάσιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις στην ε, πράξης, όταν αναφέρεται υποχρέωση για ενημέρωση, θα ήθελα να συμφωνήσω με τον εισηγητή για την ε, εμπλοκή όλων των ε, φορέων στη συζήτηση, όπως αναφέρεται στις τροπολογίες 1, 3 και 25. Και τέλος, ε, για να αποφύγουμε ένα ιδιαίτερο υπερβολικό μάλλον φόρτο, θα πρέπει υπερβολικό κόστος, θα πρέπει η υποχρέωση ενημέρωσης να επικεντρώνεται στην υπηρεσία και να μην υπάρχει επικάλυψη. Επίσης, καλωσορίζω την τροπολογία 4 του κυρίου Χατζημαρκάκη και θα ήθελα να γίνουν κάποιες ε, διευκρινήσεις σε ό,τι φορά το άρθρο 7, το Τώρα, οποιοδήποτε άλλο οργανισμό που θα έχει πρόσβαση σε αυτέ τι ευαίσθητε πληροφορίε θα πρέπει να τηρεί την υποχρέωση τη εμπιστευτικότητα του άρθρου 9. Δηλαδή αυτή η υποχρέωση πρέπει να πληρείται από όλους όσοι διαθέτουν αυτές τις πληροφορίες. Και η πληροφορία αυτή θα πρέπει να προστατεύεται και να γίνεται αυτής της πληροφορίας αποκλειστική χρήση για τους λόγους που έχουν προσδιοριστεί. Σαφώς αυτό αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Το έγγραφό του έχει μια εξαιρετική δομή και ε, συμπεριλαμβάνει όλες τις βασικές αρχές που θα διέπουν τη μελλοντική λειτουργία της ενεργειακής αγοράς. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ταχύτατα υπέβαλε το έγγραφο που θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις μελλοντικέ εξελίξεις. Ο θέμητος ανταγωνισμός στην ενεργική αγορά επηρεάζει όχι μόνο τις τιμές, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα πολιτικό μέσο μόχλευσης, ένα πολιτικό μέσο επιρροής, ας το πούμε έτσι, διότι καταβάλλονται τεράστια ποσά, διότι μέχρι στιγμής έχουμε αποτύχει στη δημιουργία μιας ενιαίας ενεργειακής αγοράς. Ε, μέχρι πρόσφατα συζητούσαμε το θέμα των τροφίμων, των ε, βασικών ζωοτροφών και καταλήξαμε στο ότι η κερδοσκοπία είναι ένα από του βασικού λόγου για του οποίου αυξάνονται οι τιμέ των τροφίμων και των ζωοτροφών σε πολλέ χώρε Το θα μπορούσε να λεχθεί και για τι ε, τιμέ των ενεργειακών προϊόντων. Θα ήθελα να σταθώ στι ε, βασικέ αρχέ του εγγράφου. Ε, επικροτώ τη σημασία που δίνεται στην αρχή της διαφάνειας, στην συγκρότηση του οργανισμού μέσα στην έκθεση του κ. Χατζημαρκάκη, χρειαζόμαστε ένα σύστημα συλλογής δεδομένων που θα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο μέλλον. Αν θέλουμε να κάνουμε μια προβολή και να φανταστούμε πώς θα διαμορφωθεί η μελλοντική μας στρατηγική, θα πρέπει αρχίζοντας να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει παντελής έλλειψη ομοιόμορφων στατιστικών ε, δεδομένων προς το παρόν. Ε, δεν υπάρχουν συγκρίσιμα εθνικά δεδομένα τα ομοιόμορφα, στατιστικά στοιχεία προφανέστατα θα είναι υποφελή για όλους μας. Δεύτερο σημείο που θα ήθελα να σχολιάσω είναι η αγορά του διοξιδίου του άνθρακος. Ε, έχω κάποιους συνδυασμούς σε σχέση με τις ε, προτάσεις που βλέπουμε στο έγγραφο. Δεν θα έπρεπε να επεκτείνουμε ανεξέλεγκτα το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Ε, και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο βασικό στόχο που είναι η δημιουργία μιας ενιαίας ενεργειακής αγοράς γιατί με την οικοδόμηση μιας τέτοιας αγοράς θα μπορέσουμε να καταλήξουμε ε, στις βασικές αρχές που θα πρέπει μελλοντικά να διέπουν την αγορά του διοξιδίου του άνθρακα στην Λιθουανία. Έχουμε ένα σαφέστατο παράδειγμα. Κλείνουμε την Ιγναλίνα που είναι ένα πυρηνικό εργοστάσιο και τώρα τελικά πληρώνουμε ακριβότερα την ενέργεια ενέργεια. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ε, παράδειγμα κατάχρησης της θέσης στην αγορά που έχει ο βασικός ε, πάροχος, βασικός φορέας εκμετάλλευσης. Για το φυσικό αέριο τώρα ε, θα αυξηθεί αναμφίβολα η ζήτηση για το φυσικό αέριο στο μέλλον, οπότε θεωρώ πως θα έπρεπε με στην έκθεση να αναφερθούμε και σε αυτό το στόχο μας, δηλαδή να δημιουργηθεί ένα όμιλο προμήθεια φυσικού αερίου που μα είχε προτείνει πέρσι ο κ. Μπούζεκ. Ε, εν γέννη, Ε, θα έλεγα ότι δοκιμάζω την έκθεση. Βέβαια θα υποβάλουμε τροπολογίες ε, έχοντας κατά νου ότι ο στόχο στόχος ε, είναι το 2014 να έχουν καταργηθεί όλοι οι ενεργειακοί νήσοι και να έχει δημιουργηθεί το νέο σύστημα παραγωγής ενέργειας που προβλέπεται στο έγγραφο. Ευχαριστώ. Ο σκιώτης συζητητής των κύριος Φόμποντα δεν ε, μπορεί να είναι παρόν εδώ πέρα. Συνεργαζόμαστε στενά. Ε, έχει συναντηθεί ήδη με τον κύριο Χατζημαρκάκη. Και βεβαίως υποστηρίζουμε πλήρως αυτά τα οποία έχει πει εδώ πέρα ο Γιώργος. Ε, μπορούμε να μιλάμε για λεπτομέρειες. Πάντα μπορεί να βελτιωθεί μια προτινόμενη νομοθεσία, αλλά κάτι στα μάτια μου νομίζω είναι ε, ξεκάθαρο είναι πως είναι απολύτως απαραίτητος ο κανονισμός. Εγώ είμαι υπέρ της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και ξέρετε πως εκεί όπου υπάρχει δύναμη υπάρχει και κατάχρηση της δύναμης ή τουλάχιστον απόπειρα να γίνει αυτό. Βεβαίως ε, υπάρχει μια σχετική οδηγία η οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν ισχύει για το τομέα της ενέργειας οπότε η Κομισιόν κατέληξε σε αυτή την πρόταση. Τώρα για το λέξη Specialis που λέει ο Γιώργος είναι απολύτως απαραίτητος κατά την απόψή μου. Πρέπει βεβαίως να ξέρουμε πως όταν μιλάμε για τα χρηματιστήρια αερίου και ρεύματος και τις σχετικές συμβάσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μιλάμε για πραγματικό ρεύμα, αλλά για κάτι το εικονικό. Και στις αγορές αυτές ε, δεν είναι μόνο άνθρωποι οι οποίοι εμπορεύονται εμπόριο και ρεύμα, αλλά τράπεζες, ε, hedge funds ε, και λοιποί εμπλεκόμενοι στην αγορά. Και καμιά φορά οι διακυμάνσεις των ε, τιμών ε, δεν μπορούν να εξηγηθούν και η γεγονός είναι πως οι απελευθερωμένες αγορές μειώνουν βεβαίω τα αποθέματα και γίνονται ακόμη πιο ακραίες οι διακυμάνσεις αυτών των τιμών. Αυτό βεβαίω είναι κάτι που χαροποιεί πάντα τους εμπόρους γιατί έτσι κερδίζουν πολύ περισσότερα και όχι με τις τιμές που ανεβαίνουν. Το 2008 παραδείγματος χάρη στις αγορές spot ρεύματος η μεγαβατόρα πήγε από 130 ευρώ σε 2.400. Μεταξύ 16 και 17 Ιανουαρίου φέτος η τιμή spot τετραπλασιάστηκε εντός λίγων ωρών από 15 στα 60 ευρώ γιατί μια μεγάλη εταιρεία αγόρασε τα πάντα, ό,τι ήταν διαθέσιμο και υπήρχε η απλή εξήγηση πως ε, ένας μεγάλος προμηθευτής θα έβγαινε από την αγορά. Χαρακτηριστική περίπτωση εσωτερικής πληροφόρησης. Ε, γι' αυτό νομίζω και βεβαίω αυτό βλάπτει καταναλωτέ και χρήστες. Γι' αυτό χρειάζεται αυτό ο κανονισμός και στην Επιτροπή Οικονομικών θα συστήσω να υιοθετήσουμε την έκθεση αυτή. Δύο παρατηρήσει τρει ακόμα. Εάν ε, γίνει δεκτός αυτός ο οργανισμός, βεβαίως θα πρέπει η υπηρεσία αυτή, η Acer, η οποία λειτουργεί στη Λουμπλιάνα εδώ και κάτι εβδομάδες, να λάβει χρηματοδότηση. Χωρίς λεφτά δεν θα μπορέσει να κάνει αυτή την επιπρόσθετη εργασία. Τώρα για τα προβλήματα που ανέφερε ο Γιώργος Χατζημαρκάκης, δηλαδή για την επέκταση και στην αγορά του διοξιδίου του άνθρακα. Επί της αρχής είμαι υπέρ γιατί ζήσαμε πόσο ακριβώς στις αγορές του οξύδου του άνθρακα είχαμε και επιθέσεις ηλεκτρονικές αλλά και απάτες σε πολύ μεγάλο ύψος. Αναμένουμε λοιπόν τοποθέτηση από την Κομισιόν επί της πρότασης Χάτζη Μαρκάκη η αντιπρόταση που θα μπορούσε να μας ικανοποίηση. Η Κομισιόν ανέφερε πως θα κάνει νέα διατύπωση της οδηγίας BFID και βελτίωσή της και φανταζόμαστε πως το εμπόριο διοξιδίου του άνθρακα θα καλύπτεται είτε σε αυτό το πλαίσιο είτε σε ένα λέξη σπεσιάλης αλλά δεν μπορούμε να αποδεχτούμε το εμπόριο διοξιδίου του άνθρακα να αποτελεί πεδίο δράσης απαταιώνων και κερδοσκόπων. Όταν μιλάμε επίσης για κανόνες, μιλάμε και για κυρώσεις. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, να οδηγηθούμε δηλαδή σε μια εναρμόνιση των κυρώσεων. Ένα συνάλφος του ΕΛΚ παρατήρησε πως κανονικά Δεν το θέλουν αυτό τα κράτη-μέλη γιατί λένε εμείς είμαστε υπεύθυνα για τις κυρώσεις. Οπότε θα μπορούσαν βεβαίως να αποφασίζουν για τις κυρώσεις αλλά για να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού οι κυρώσεις θα μπορούσαν να είναι βεβαίως αποτελεσματικές και να έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα. Και εδώ πέρα βεβαίω στηρίζουμε πλήρω τον κύριο Χάτζη Μαρκάκη. Ευχαριστώ, επειδή όμω θα έρθει και ο Επίτροπο, να δώσω τον λόγο στην Κομισιόν για δύο-τρία λεπτάκια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Χάτζη Μαρκάκη και τους υπόλοιπους ομιλητές γιατί νομίζω πως ήταν θετικά, θετική η σημερινή συζήτηση τους ευχαριστούμε και τον εισηγητή για τη συνεργασία. Είμαστε ευγνώμονες για τη στήριξή του. Ε, δεν θα τονίσω τώρα που συμφωνούμε. Αναφερθώ στα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν εδώ. και ο κύριος Γκέμπελς και άλλοι ανέφεραν το θέμα του διοξείδου του άνθρακα. Τους διαβεβαιώ πως η Κομισιόν δεν θέλει να γίνεται αυτό το εμπόριο σε έναν χώρο εκτός νόμου. Πρέπει να ρυθμιστεί. Οπότε το εμπόριο διοξιδίου του ανθράκα καλύπτεται καλύτερα από το MIFID παρά από την οδηγία. μείτε εδώ. Κατ' ουσίαν πρόκειται για τα χρηματοοικονομικά μέσα και οι ρυθμιστικές αρχές αυτές άρα είναι καλύτερες για να το ελέγξουν αυτό το θέμα. Θα ήμασταν όμως ανοιχτοί στο να δει αυτό το εμπόριο διοξιδίου του ανθρακά και η Acer όσον αφορά τις αρμόδιες αρχές και ποιες είναι. Και το ιδιαίτερο πρόβλημα της Γερμανίας περί σύστασης υπηρεσίας διαφάνειας. Εμείς ε, συμφωνούμε με τον κύριο Τούρμες. Δεν ε, πρέπει να δημιουργήσουμε ψηφιδωτό εδώ πέρα, μοσαϊκό. Οι αρχές αυτές πρέπει να αποτελέσουν την ε, ραχοκοκαλιά της Acer. Θα πρέπει να συνεργάζονται με συναδέλφους τους, άρα ε, στο ρυθμιστικό συμβούλιο της Acer, δηλαδή τις εποπτικές αρχές για την ενέργεια και θεωρούμε πως ε, δεν χρειάζεται, όπως υπόθηκε πάλι άλλο ένα μοσαϊκό. Οι αρχές εποπτείας ενέργειας είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να είναι σε επαφή και να ασκούν την εποπτεία. Για το θέμα των πράξεων κατά εξουσιοδότηση, αυτό εμφανίζεται μόνο σε δύο σημεία στην πρότασή μας. Θεωρούμε πως η Κομισιόν όσον αφορά την ενημέρωση των ορισμών Όταν ε, ήταν κάτι παράλογο με, αυτό, με κάτι με αυτό το οποίο είχαμε κάνει και για το short selling. Οπότε νομίζω πως είναι το κατάλληλο μέσο για αυτές τις αποφάσεις. Όσον αφορά την αδειοδότηση, είμαστε κάπως πιο επιφυλακτικοί από τον κύριο Χατζή Μαρκάκη. Και βεβαίως ως μια θέση αναδίπλωσης θα μπορούσαμε να σκεφτούμε την καταγραφή. Αλλά για διοδότηση θεωρούμε πως δεν υπάρχει λόγος. Όσον αφορά τις κυρώσεις, αναφέρθηκαν ήδη πολλά επιχειρήματα, μπορούσαμε να δούμε τι γίνεται με τις ε, υπόλοιπες αγορές για να βρούμε μία λύση για τον τομέα ρεύματος και αερίου. Για τις αγορές εκτός Ένωσης, η Νορβηγία είπατε σωστά δεν είναι πρόβλημα. Η συμπερίληψη της ελβετικής αγοράς θα είναι δύσκολη. Εκτός αν βρούμε λύσεις στις διμερείς διαπραγματεύσεις. Απλά να σας πω πως οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δεν, ε, που δεν δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης πρέπει ούτως ή άλλως να τα δηλώνουν αυτά στην Ελβετία. Δεν έκανα μαύρο κουτί δηλαδή που χάνονται εκεί μέσα. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Όσον αφορά τη δυνατότητα γραφείων εκπροσώπησης της Acer σε διάφορες πόλεις Ευρώπης, και εγώ είμαι επιφυλακτικό. Εντάξει, να έχει ένα γραφείο εδώ στι Βρυξέλλε, αλλά τώρα σήμερα στον καιρό τη τεχνολογία δεν χρειαζόμαστε και άλλα γραφεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οπότε δεν χρειάζεται ε, άλλη γραφειοκρατία. Η πρόταση του κυρίου Τούρμες περί περιφερειακών αγορών είναι ενδιαφέρουσα. Και τελειώνω κύριε Πρόεδρε και οι υπόλοιπε παρατηρήσει του κυρίου Βιδάλ Κουάντρα πρέπει να τις δούμε. Είναι ενδιαφέρουσε. αλλά εξαρτάται από το πώ θα διατυπωθούν. Ευχαριστώ και τον κύριο Χατζημαρκάκη και όλους σας για την θετική αντιμετώπιση της πρότασης μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χατζημαρκάκης πάλι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Κομισιόν που αναφέρθηκε σε όλα τα σημεία. Νομίζω θα βρούμε κανένα συμβασμό για τα γραφεία συνδέσμου. Δεν θέλουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη να ανοίξουμε γραφεία σε ένα-δύο σημεία εμπορίας. Όχι μόνο για να υπάρχει άμεση εικόνα, αλλά και για να δημιουργήσουμε ελκυστικές δουλειές. Ξέρετε, γιατί δεν πάει εύκολα ο κόσμος στη Λιουμπλιάνα. Δεν είναι συγκρίσιμα τα πράγματα με τη ΣΥΠΑ. Δηλαδή, το να πάει ένας Ισπανός Σλοβενία έχει πρόβλημα να πάει τα παιδιά του στο σχολείο στις Βρυξέλλες στο Παρίσι είναι απλούστερο. Με αυτό είναι σημαντικό το γραφείο αυτό συνδέσμου. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους. Σας ευχαριστώ. 19 Απριλίου, 12 η ώρα προθυμία για τροπολογίες. Τελειώσαμε το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Διαλυματάκι, να σας υπενθυμίσω πως στην έκθεση Τσίτσεστερ η προθεσμία είναι 13 Τετάρτου για τις τροπολογίες. Και περνάμε στο επόμενο σημείο, την επίσκεψη του κυρίου Έτσιγκερ, εδώ είναι ήδη. Τον καλωσορίζω.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 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας πω τι θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες και βεβαίως τα βασικότερα πράγματα που είναι σημαντικά για την Κομισιόν στο κλίμα και την ενέργεια. Ξεκινώντας από το Συμβούλιο της 4ης ε, ε, Φεβρουαρίου, θα εκμεταλλευτούμε τις οθήσεις που δόθηκαν εκεί για να προωθηθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν 15 χρόνια μετά την νομοθέτηση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας να μην υπάρχει αυτή στην πραγματικότητα. Υπάρχουν με μεμονωμένες αγορές, δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Ναι, τα κράτη-μέλη μάλιστα θεωρούν ακόμη περισσότερο πως θα πρέπει να προστατεύουν και να επιδοτούν τις δικές τους επιχειρήσεις. Οπότε, αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε τη διαδικασία για την εφαρμογή του τρίτου πακέτου εσωτερικής αγοράς πρέπει να έχει ήδη εφαρμοστεί μέχρι το καλοκαίρι θα παρακολουθούμε τη διαδικασία και μετά το δεύτερο εξάμεινο εκεί όπου δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως η εσωτερική αγορά θα κινηθούμε αναλόγως. Δεύτερον, θέλουμε να φέρουμε στο προσκήνιο την εξωτερική διάσταση και να γίνει μια ανακοίνωση για μια εξωτερική πολιτική ενέργεια της Ένωσης. Θα υπάρξει λοιπόν μια ανακοίνωση από πλευράς Κομισιόν και Συμβουλίου και θα δούμε μαζί το θέμα του πού έχει νόημα μια τέτοια πολιτική. Δεν θα αντικαταστήσει την πολιτική των κρατών μελών, αλλά θα την συμπληρώσει εκεί όπου ε, θα έχουμε να επιτύχουμε ευρωπαϊκούς ενεργειακούς στόχους και εκεί όπου είναι καλύτερο να οργανωθούμε από κοινού. Δηλαδή στο θέμα Ανατολική Ευρώπη, Νότιο Ανατολική Ευρώπη, Κασπία και Μεσόγειος. Εκεί μου φαίνεται πως ε, θα πρέπει να έχουμε μια κοινή εξωτερική πολιτική. Τρίτον, από Μάιο θα προετοιμάσουμε τον ενεργειακό δικό χάρτη 2050 κάτι το φιλόδοξο σκεφτείτε λίγο τι γινόταν στο 1970 εάν κοίταγε κανείς το 2011 τι θα πριν ε, γνωρίζει κανείς βεβαίως ε, την πετρελαϊκή κρίση, την πτώση του τείχους, τις, ε, τις επιστημονικές αλλαγές, πώς μπορούσε να προβλέψει το 2011. Εξίσου δύσκολο είναι να προβλέψουμε το 2050, αλλά το θέμα δεν είναι η ημερομηνία, το θέμα είναι πώς θα αλλάξει το ενεργειακό τοπίο 2025-2030 και μέχρι το 2040, γιατί οι επενδυτές ανεξαρτήτως των ανεπενδύων επενδύουν στην παραγωγή, στην αποθήκευση, στην έρευνα ή στην υποδομή, χρειάζονται ασφάλεια για τον προγραμματισμό τους. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει αυτή η ασφάλεια για τους επενδυτές για να μπορέσουμε περισσότερο από τη τώρα να προσελκύσουμε επενδυτικές ροές στην ενέργεια. Προετοιμάζουμε επίσης τα τεστ κοπόσεως. Σημαντικό αυτό για το έργο μας το 2011. Είμαστε σε επαφή με τις Εθνικές Υπηρεσίες Ατομικής Ενέργειας για τα κριτήρια εξέτασης για να αποφασίσουμε ποιος θα εξεταστεί Και όλα αυτά βεβαίως με το στόχο να μπορέσουμε να υποβάλουμε τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου στο Συμβούλιο που θα γίνει τα Χριστούγεννα. Και αυτή τη στιγμή κάνουμε αυτές τις ε, συζητήσεις ή γίνεται αυτή η ε, εξέταση λοιπόν για να δούμε πώς θα γίνουν τέσσερα ποσό είμαστε σε επαφή με την Ουκρανία, με τη Ρωσία, την επόμενη εβδομάδα με την Ελβετία. Έχουμε αποστείλει προσκλήσεις στην Αρμενία και την Κροατία αλλά και χώρες που δεν έχουν ακόμα πυρηνικά εργοστάσια όπως η Τουρκία και η Λευκορωσία ε, θα κάνουν ένα τέτοιο έλεγχο. Τους έχουμε ζητήσει να ενταχθούν σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Επίσης, μετά την πρώτη μας ανακοίνωση. Θα επανεπεξεργαστούμε τις οδηγίες TEN E, ε, και τα της χρηματοδότησης. Το θέμα δε των υποδομών πρέπει να αποκτήσει μεγάλη σημασία. Επίσης έχουμε και τα μέτρα αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας με στόχο 20% σε 9 χρόνια με μια διπλή στρατηγική. Αυτή τη στιγμή εθελοντικά, αλλά κάποια μέτρα θα γίνουν υποχρεωτικά και το αργότερο από το 2013-2014 με δεσμευτικούς στόχους αν δεν ε, υπάρχει πρόοδος. Στα δημόσια κτίρια αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία για να κινητοποιήσουμε την αγορά, για να παίξουν ρόλο προτύπου, αλλά και γιατί ο δημόσιος τομέας έχει το 12% όλων των κτηρίων. Σχολεία, πανεπιστήμια, κοινοβούλια, στρατώνες, δημαρχία, γυροκομεία. Και βεβαίω υπάρχει και το ζήτημα της ενεργειακής αποτελεσματικότητα. Μιλάμε ε, για μια επένδυση μόνο 1,5% το έτος. Με αυτό το στόχο βεβαίω θα χρειαστούν ε, πάρα πολλά χρόνια. Επειδή όμως η τεχνολογία ανανεώνεται πάρα πολύ γρήγορα πρέπει να φτάσουμε σε ένα επίπεδο επένδυσης 3% και βεβαίως ε, θα πρέπει όπως σας είπα ένα 3% των δημοσίων κτηρίων να έχουν γίνει ενεργειακά αποτελεσματικότερα και βεβαίω θα πρέπει να το δούμε αυτό και από πλευρά ευρωπαϊκού προπολογισμού, ταμείων συνοχής κτλ. Γιατί βεβαίω δεν μπορεί να τα κάνουν αυτά 100% ε, τα κράτη-μέλη. Γιατί εγώ θέλω ήδη στον ορεινό προϋπολογισμό αλλά και από τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές να αποτελέσει προτεραιότητα των διαρθρωτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην έχετε ψευδεστήσεις. Στα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει πάρα πολλά στα κτίρια, αλλά κυρίως μιλάμε για γύψο, αν θέλετε, δηλαδή για α, ανακαινήσεις Ανακαινήσεις όμως όχι ενεργειακές. Οι ενεργειακές ε, ανακαινήσεις είναι αόρατες. Δεν βλέπουμε μετά κάτι το ωραίο. Και μιλάμε για 500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Και Νομίζω πω θα παίξει εδώ πέρα, άρα οι υποχρεωτικές διατάξει για το δημόσιο τομέα θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Μετά, το θέμα έξυπνα δικτύα. είναι λοιπόν πάρα πολύ μεγάλο θέμα να έχουμε δίκτυα, γιατί ξέρετε θα έχουμε τις ε, θαλάσσιες εγκαταστάσεις στη Βόρεια Θάλασσα που θα πρέπει να τροφοδοτούν τις Μετροπόλεις της Ευρώπης και έξυπνα ρολόγια, έξυπνους μετρητές για την κατανάλωση. Δεν πρέπει να τα υποτιμούμε αυτά. Οπότε η ανακοίνωση περί έξυπνων δικτύων είναι πάρα πολύ σημαντική. Μιλάμε για ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών, μιλάμε βεβαίως για ζητήματα προστασίας δεδομένων των καταναλωτών, για ένα νομικό πλαίσιο για να έχουμε τα έξυπνα δίκτυα αυτά, έρευνα και ανάπτυξη και νέα συστήματα και άρα το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Και μετά γενικά για την έρευνα, με τη συνάλφο Γκέγγεν Κουίν έχουμε μια καλή επαφή και από τις 4 ε, Μαΐου τουλάχιστον θα πρέπει να δούμε δύο θέματα όσον αφορά την ενεργειακή έρευνα. Τεχνολογίες δικτύων και τεχνολογίες αποθήκευσης. Γιατί πέρα από τον υδροηλεκτρικό τομέα δεν έχουμε τίποτα όσον αφορά την αποθήκευση και δεν έχουμε νέες τεχνολογίες αποθήκευσης ρεύματος. Αν μου επιτρέπετε να χαράξω ένα όραμα. Πριν από έξι μήνες είχαμε την οδηγία για το φυσικό αέριο και αποφασίσατε πως θα πρέπει να υπάρχει φυσικό αέριο από θέματα 30 ημερών έτσι ώστε να μην βρεθεί σε έσχατη ανάγκη και να μην ε, πέσει η ποιότητα ζωής ε, και θέρμανση κτλ. Οπότε θέλω να έχουμε και αποθηκευμένο ρεύμα για 30 ημέρες ως υποχρεωτική οδηγία. Βεβαίως αυτό στη στιγμή κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο, αλλά θα μπορούσαμε με οξυγόνο, με πεπιεσμένο αέρα, με μπαταρίες. Δεν θεωρώ πως είναι κάτι το αδιανόητο. Äh, Μετά έχουμε υπερακτιο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, να δούμε ποια είναι τα παραθυράκια εκεί πέρα στην νομοθεσία και να καταλήξουμε σε ευρωπαϊκές διατάξεις. Αυτά νομίζω είναι τα βασικά σημεία τα οποία θα ολοκληρωθούν στη διάρκεια του έτους ή θα ξεκινήσουν. Και βεβαίως ευχαρίστως διμερός με την Επιτροπή σας να ε, είμαστε σε επαφή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχουμε μέχρι τις 5 ε, χρόνο να σας ακούσουμε. Οπότε, να αφήσουμε έτσι τους χαιρετισμού και να λέμε πόσο ωραίος είναι ο Επίτροπος και τέτοια, να περάσουμε κατευθείαν σε ερωτήσεις. Εντάξει, ξέρουμε όλοι, τον ευχαριστούμε που ήρθε μείνετε σε ερωτήσεις για να πιέσουμε τον Επίτροπο να πει και συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, δύο λεπτά παρακαλώ. Κυρία Αντελκαστήγια. Ναι, συγχαρητήρια ούτω ή άλλω. Τώρα θα αναφερθώ στα σημεία που μα ενδιαφέρουν περισσότερο. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση, η οποία ήταν πληρέστατη σχετικά με τα θέματα της ενέργειας. Τώρα, Επίτροπε, αναφερθήκατε στην ε, δυνατότητα μιας εξωτερικής πολιτικής ενέργειας σε ορισμένα ζητήματα. Αυτή η πρωτοβουλία θα αναπτυχθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όμως την Ήτρε και να μην ε, βρεθεί βρεθούμε στην κατάσταση η Επιτροπή Εξωτερικών να είναι αυτή που θα εξετάσει και θα αναλύσει αυτή τη νέα διάσταση. Για μα είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, δεν πρέπει να ξεχάσετε. Τώρα, να αυτό το εξή. Προημερών στο Στρασβούργο υπήρξε ένα κοινό ψήφισμα σχετικά με την καταστροφή μετά από το τσουνάμι, τον σεισμό κλπ. της Ιαπωνίας, στον σταθμό της Φουκουσίμα και το ψήφισμα τελικά δεν εγκρίθηκε στην ψηφοφορία. Αλλά ορισμένα από τα σημεία που περιέχονται στην ε, ψήφισμα ε, χρησιμεύουν στην Κομισιόν για να γνωρίζει τη θέση του Κοινοβουλίου επί συγκεκριμένων και πολύ σημαντικών θεμάτων. Πρώτα απ' όλα, πώς ε, χρειάζεται να γίνει μια σειρά από τεστ ε, τεστ αντοχής ε, στους πυρηνικούς σταθμούς και το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι αυτές οι δοκιμές πρέπει να είναι υποχρεωτικές και με βάση κοινά κριτήρια και την ε, η ηγεσία αυτών των τεστ θα πρέπει να ανελθεί από την Ευρωπαϊκή Τροπή. Θα χρειαστεί φυσικά να γίνουν δοκιμές και σε γειτονικέ χώρες αλλά και σε χώρες που κατασκευάζουν πυρηνικούς σταθμούς. Τώρα η πυρηνική ενέργεια είναι κάτι που ε, είναι απαραίτητο σήμερα. Δεν θέλω να πούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ως εκ τούτου είναι ένα ζήτημα σαφές για το Κοινοβούλιο ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πέραν του 20% μετά το 2020 δεν θεωρείται ως ρεαλιστικό για να επιτευχθεί και τέλος θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα ITER θα πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτείται διότι κρίνουμε ότι είναι ένα σημαντικότατο πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το μέλλον της ενέργειας πανταχού στον κόσμο. Ευχαριστώ. Μπομπίνσκα. Ευχαριστώ. Το ίδιο στοιχείο θα ήθελα να σχολιάσω. Ξέρετε ότι επέτυχε το, η πρόταση κοινού ψηφίσματος στο Στρασβούργο για τη Φουκουσίμα και τα θέματα ασφαλείας στα πλαίσια τη ενεργειακής πολιτικής. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή. Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα προς επίρρωση της ευρωπαϊκής πολιτικής ε, για την ε, πυρηνική ασφάλεια. Μας μιλήσατε για τα τεστ κοπόσεως, τα τεστ αντοχής, αλλά μετά από αυτά τι θα γίνει, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Το σημείο καμπής θα είναι η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει. Και πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι επί πολωνικής προεδρίας ή αργότερα. Τώρα για τη χρηματοδότηση των υποδομών θα ήθελα να στέσω και άλλη μια ερώτηση. Έχετε κάποια ιδέα σχετικά με τα μέσα, τα εργαλεία που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε για να κατοχυρώσουμε τη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να έχουμε ένα ξεχωριστό μέσο ή μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε μέσα το, της διαρθρωτικής ε, πολιτικής. Και τι πιστεύετε για τη διαφοροποίηση των χρηματοδοτικών ε, μέσων εν Ευχαριστώ. Μπέλετ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, άκουσα. Διάβασα την ε, συνέντευξή σας στο Σπίγγελ και προκύπτει από εκεί πως θέλετε να πάμε προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υπάρχουν βεβαίως κάποιες βασικές προκλήσεις. Αναφέρατε αποθήκευση της ενέργειας, μπαταρίες κτλ. Το άλλο, υποδομές, οι αυτοκινητόδρομοι αν θέλετε ανανεώσιμης ενέργειας από βορρά προς νότο και ανατολή προς δύση και το επόμενο σημείο στην για διαταξή μας βεβαίως το θέμα της κυρίας Σόζα Βάγνερ και βεβαίως ξέρετε πως ε, θα έχουμε πάρα πολλές ε, αντιδράσεις και καθυστερήσεις από τους ε, πολίτες. Οπότε ποιες είναι οι δυνατότητες ε, να έχουμε πιλωτικά ε, έργα για να είναι υπόγεια αυτά τα έργα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τέλος όσον αφορά τα οικονομικά μέσα πέρα από τα ευρωομόλογα το πώς θα μπορούσαμε π.χ ένα μεγάλο κομμάτι των ε, κερδών ε, των πυρηνικών εργοστασίων να πάνε σε ε, επενδύσεις στην ανανεώσιμη ενέργεια. Τι άποψη έχετε αυτό. Η κυρία Τζαβέλα. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας κάνω τρεις ερωτήσεις σχετικά με την χρηματοδότηση των υποδομών. πολύ ελκυστικό μέσο φαίνεται να είναι τα project bonds, τα οποία θα μπορέσουν να αντλήσουν κεφάλαια για τις υποδομές στην ενέργεια από τον ιδιωτικό τομέα. Η Επιτροπή προβλέπει λειτουργία αυτού του, της πρωτοβουλίας το 2014. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ αργά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με αυτό το μηχανισμό χρηματοδότησης. Θα μπορούσατε να δείτε αν μπορούμε πιο γρήγορα, τουλάχιστον για την ενέργεια, να προχωρήσουμε στα project bonds για να χρηματοδοτήσουμε υποδομές. Για την αλλαγή του ενεργειακού τοπίου, έχετε σχεδιάσει ή σχεδιάζετε ή κάνετε απογραφή των ιδίων πηγών ενέργειας, προμήθειας ενέργειας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας έχουμε και το γκάζ λένε ότι στο νότο στη Μεσόγειο υπάρχουν αποθέματα αερίου τόσα όσα έχει το ΣΑΧΔΕΝΗΣ. Ε, έχετε καταγράψει το θέμα του shale gas. Οι Αμερικανοί αναφέρουν ότι η Γερμανία διαθέτει 8-3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα shale gas στο έδαφος της. Άρα λοιπόν η Ευρώπη έχει ίδιους πόρους επ' αυτού του θέματος. Μπορούμε να κάνουμε μια καταγραφή για να δούμε τι έχουμε. Και το τρίτο και τελευταίο, αναφερθήκατε στα, τεστ, στα stress test των πυρηνικών μονάδων, δεν είπατε για τη Ρουμανία όπου έχουμε το εργοστάσιο Τσερναβόντα από το 1980 που θα ξεκινήσει με τρεις αντιδραστήρες. Ευχαριστώ. Kollegin Niebler. Νίμπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε. Τρεις παρατηρήσεις. Να αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπε η κυρία Πιλάρντε Καστίγιο και η κυρία Κολάρσκα. Ο Μινσκά. Ήμουν εδώ την προηγούμενη εβδομάδα σε ολόκληρη την συζήτηση και ε, και δεν εγκρίθηκε το ψήφισμα περί Φουκουσίμα, όλοι είπαν πως θα πρέπει να έχουμε τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας για τα εργοστάσια για τα πυρηνικά στην Ευρώπη. Νομίζω πως αυτό είναι το πολιτικό μήνυμα του Κοινοβουλίου, αν και δεν καταλήξαμε σε κάποιο ψήφισμα. Δεύτερον, Μιλήσατε για τον ενεργειακό χάρτη 2050, την εξωτερική διάσταση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω εδώ πέρα το Desert το έργο στην ε, Βόρεια Αφρική, για να εξυπηρετήσουμε και την Ευρώπη. Θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκό έργο και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύει να λάβει η ε, Κομισιόν για να προωθήσει το Desert Tech. Και τέλος, παλιό θέμα, ξεκινήσατε με την εσωτερική αγορά της ενέργειας, είπατε πως δεν υπάρχει τέτοια, γιατί υπάρχει προσταταυτισμός και εθνική αγορά και σας παρακαλώ να μην δώσετε μόνο βάρος στις ιδιωτικές εταιρείες, υπάρχουν και κρατικά μονοπόλια σε πολλές ε, χώρες. Και αν κάνετε κάτι με αυτό θα είχατε τη στήριξη πολλών στην Επιτροπή μας. Κύριε Καρβάλιο, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Συγχαίρω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρωτευουλία για τις διεθνούς διάστασεις στον τομέα της ενέργειας θα συμφωνήσω με τη συνάδελφο Καστίγιο ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή για το ζήτημα αυτό. Ήθελα να αναφερθώ μόνο στη σημασία του Ατλαντικού μετώπου. Ε, στα πλαίσια της ε, διεθνούς διάστασης και στο Βορρά και στο Νότο. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ακτές της Δυτικής Αφρικής έχει ξανόμενη σημασία για την Ευρώπη. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι η έρευνα και χαίρομαι που σας άκουσα να λέτε πως θέλετε να αυξήσετε σημαντικά ε, τα κονδύλια για την έρευνα. Αυτή έχει κυρία σημασία διότι Χρειάζεστε προγράμματα επίδειξης και πιλωτικά προγράμματα σε πολλές περιπτώσεις στην έρευνα και δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσο σημαντική είναι η πιλωτική κλίμακα και η επίδειξη για, την, ε, για το για την επόμενη γενιά ερευνητικών προγραμμάτων. Τελευταία ερώτηση. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίε ε, σχετικά με την ανάπτυξη των προγραμμάτων επίδειξης, ε, τα προγράμματα CCS ε, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΒΡΙΚΑ γιατί έχουν αντιμετωπίσει ε, κάποια προβλήματα και θα ήθελα, αν μπορείτε να μας ενημερώσετε για την εξέλιξη αυτών των προγραμμάτων. Ευχαριστούμε. Για να ξεκαθαρίσω τώρα τη σειρά των ε, ομιλητών, θα πω τα ονόματα και ε, παρακαλώ να μην καθυστερείτε. Ναι, το με τη σειρά λοιπόν όσοι ζήτησαν το λόγο θα πάρουν το λόγο εκτός αν θέλουν οι ίδιες πολιτικές ομάδες να αλλάξουν τη σειρά. Ο κύριος Γκέμπελ. Έχουμε την πρόταση της Κομισιόν ε, για έναν οδικό χάρτη για το 2050. Αυτό είναι αφηρημένο. Δεν είναι δυνατόν τώρα να ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι το 2050 θα είναι φαντασίες και ευσεβείς πόθη, αλλά στην πραγματικότητα δεν εξυπηρετούν τίποτα. Είπατε και ο ίδιος πως η τεχνολογία ε, κάθε 20 χρόνια ανανεώνεται εκ Δηλαδή δύο φορές θα έχουν περάσει 20 χρόνια μέχρι το 2050. η Κομισιόν σκέφτεται πάρα πολλά τέτοια πράγματα αυτή τη στιγμή βέβαια για το 2050, αλλά 2050 από τους παρόντες δεν θα είναι εδώ κανείς. Γιατί βεβαίως ε, μην ξεχνάμε πως ε, ε, παίρνουμε και διάφορες αποφάσεις και λέμε 50%, ε, 100% ε, ξέρω εγώ των, ε, της ενέργειας θα είναι, από ανανεώσιμες πηγές. Π.χ. με τη Φουκουσίμα φοβόμαστε την πυρηνική. Εάν αύριο έχουμε έκρηξη σε ένα τάνκερ μεθανίου, θα έχουμε πάλι εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες θύματα, που δεν το ελπίζω. Και θα αλλάξει ξανά η ενεργειακή πολιτική. Μπορώ να αναφέρω και άλλα τέτοια παραδείγματα. Η ΔΕ Γερμανία μετά τη Φουκουσίμα αποφάσισε να κλείσει κάποια τέτοια εργοστάσια. Αλλά έκτοτε από εξαγωγέας έγινε εισαγωγέας ε, ηλεκτρικού ρεύματος με μεγάλα προβλήματα για την υπόλοιπη Ευρώπη. Και ανησυχώ για το τι θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι εάν ε, έχουμε στενοπούς αν θέλετε, στην παροχή ρεύματος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οπότε εσείς και η υπηρεσία σας θα πρέπει να επικεντρωθείτε στο αύριο και στο μεθαύριο. Θα ήθελα λοιπόν να τα γνωρίζω η ΑΠΕ που λέτε πώς θα μεταφορθούν, ε, πώς θα έχουμε δικτύα διασυνοριακά. Τι γίνεται με την αποθήκευση επίσης. Και αν μου επιτρέπει ο πρόεδρος, θα έχουμε μια νέα αγορά ενέργειας. Πώς θα είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά που επιθυμείτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να, σας, ε, να συγχαρώ τον Επίτροπο για την εφαρμογή του τρίτου ενεργειακού πακέτου. Πιστεύω ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ την ε, Γερμανία. Μιλήσατε για την ενεργειακή απόδοση. Όντως, ε, πολλά κράτη-μέλη δεν ε, μπόρεσαν να εφαρμόσουν τα διάφορα μέτρα των διαδοχικών πακέτων. Επί σειρά ετών παρατηρείται αυτό το φαινόμενο και νομίζω ότι πρέπει να αυξήσει την πολιτική πίεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ούτω ώστε να ακολουθούνται οι κατευθυντήριες γραμμές από όλα τα κράτη-μέλη. Ε, αναφερθήκατε στο 2014 για την έναρξη εφαρμογής του νέου προγράμματος περί εξωτερικής διάστασης. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς ακριβώς θα εφαρμόσετε την πολιτική της αντίστροφης ροής, reverse flow. Ένα άλλο θέμα σχετίζεται με την οδηγία για, την, ε, για τα αποθέματα φυσικού αερίου. Ε, μας είπατε ότι θα πρέπει να έχουμε αποθέματα για 30 ημέρες. Ε, μα αυτό απαιτεί πάρα πολύ ψηλά ποσά δεν πιστεύετε ότι η Επιτροπή για την Προμήθεια σε Φυσικό Αέριο, στην οποία αναφέρθηκε και ο Πρόεδρός μας, θα έπρεπε να εμπλακεί στο πρόγραμμα αυτό. Εν τη αυτή περίπτωση για την προμήθεια φυσικού αερίου, διότι προς το παρόν είναι αρκετά διχασμένα τα κράτη-μέλη και μονομερώς κινούνται για να προμηθευτούν φυσικό αέριο ε, και ε, τρίτες χώρες εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και νομίζω πρέπει να αναθεωρήσουμε την γραμμή που ακολουθούμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπιτικόφε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Επίτροπο για αλλαγή. Ε, τον συγχαίρω διότι ε, είχε θέσει διάφορους ε, φιλόδοξους στόχους ε, για την ενεργειακή αγορά και μόνο γι' αυτό πρέπει να το αποδώσουμε εύσημα. Τώρα τι θα γίνει με τους στόχους θα το δείξει το μέλλον. Θα ήθελα ε, να διορθώσω κάτι που είπατε. Εμείς ε, στη Γερμανία θα συνεχίσουμε να εξάγουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορεί κάποιο να ισχυριστεί το αντίθετο, αλλά πάντως τα γεγονότα παραμένουν γεγονότα και δεν μπορείτε να τα αμφισβητήσετε. Δεν ε, μπορώ παρά να εστιχηματίσω υπέρ αυτού. Θα ήθελα να περάσω σε κάποιες ερωτήσεις, κύριε Τίνκερε, για την παρουσίαση που μας κάνατε. Πέρα από αυτά τα τεστ ε, κοπόσεως, θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε το εξής. Ο τρόπος ε, αποθήκευση, προσωρινής αποθήκευσης των πυρηνικών αποβλήτων ε, στη Φουκουσίμα οδήγησε σε πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους. Οπότε δεν χρειαζόμαστε τεστ κοπόσεως, χρειαζόμαστε ξηρά αποθήκευση των αποβλήτων, ε, ξηρά προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποτρέψουμε την εξαγωγή πυρηνικών αποβλήτων. Ε, σχετικά με την εξοικονόμηση τώρα της ενέργειας, το πρόγραμμα που έχετε εκφωνήσει ενεργειακή απόδοση, θα έλεγα το εξής. Γνωρίζετε τις προθέσεις των ΜΕΡ και των ΔΕ και χρειαζόμαστε νομοθετικές προτάσεις πριν το καλοκαίρι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. ούτω ώστε σε κάποια επερχόμενη προεδρία να μπορούμε να ελπίζουμε σε μια συμφωνία για αυτόν τον ενεργειακό οδικό χάρτη. Ε, εσείς στο δικό σας σενάριο βασιζόσαστε σε ποσοστά ε, ε εικονικά 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, συμμερίζομαι τις επιθυμίες σας, ε, αλλά θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. θα πρέπει να κινηθούμε ε, ούτως ώστε να μην ε, καταναλώσουμε όλα τα κονδύνια για το ίτερε και να αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα στην, ε, στην άκρη. Κυρία Τικάου τώρα, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Το 2020 μόνο 1% των κτηρίων θα είναι νέα κτίρια. 99% των κτηρίων θα είναι παλιά κτίρια λοιπόν. Άρα η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων καταλαβαίνετε ότι αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Στην οδηγία ε, δίνουμε έμφαση στις επενδύσεις ε, που πρέπει να γίνουν για τη στέγη. Τώρα ε, για τους δημόσιους οργανισμούς, για τους δημόσιους φορείς, ε, είπαμε ότι από το 2019 και μετά η ενεργειακή κατανάλωση αυτών των κτηρίων πρέπει να κυμαίνεται σε μηδενικά ποσοστά. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα έχουμε στο μεταξύ αναλάβει τα κατάλληλα μέτρα, ούτω ώστε τα τεχνικά συστήματα των κτηρίων ε, να εγκαταστούν αποτελεσματικά από ενεργειακής άποψης. Το 2008 22 κράτη-μέλη δεν είχαν εφαρμόσει ε, την οδηγία του 2002. Πώς έχει λοιπόν η κατάσταση σήμερα. Είπατε ότι θα κάνουμε περαιτέρω επενδύσεις από το 2014 και μετά για την ενεργειακή απόδοση και ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, τα διαθέσιμα κονδύλια σε ποσοστό 100%. Μα το 100% συνυπολογίστε και τα κτίρια, διότι προς το παρόν υπάρχει ένα κατόφλι 4% για την ενεργειακή απόδοση των κτίριων. Το 2020 Ξαναλέω, 99% των κτηρίων θα είναι παλιά ε, και πρέπει να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό το θέμα. Επίσης, τίθεται ένα ε, μεθοδολογικό ζήτημα. Πώς υπολογίζονται ε, τα πρότυπα σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, η μεθοδολογία που προβλέπεται στην οδηγία του 2002 είναι εφαρμόσιμη, το χρονοδιάγρημα, είναι εφικτό. Ε, στο μέτρο που έδωσε τη σύμφωνη γνώμη το Κοινοβουλίο για τι πράξει κατά εξουσιοδότηση. Κοιτάξτε, έχουμε ακόμη 10 ομιλητέ. Δεν γίνεται να το πάρουμε ε, ε, μαθηματικά το θέμα. Δεν γίνεται, αλλά παρακαλώ να είστε όλοι σύντομοι. Κύριε Μαρίζα Ματία, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ωραία, θα υπακούσω ευθύ αμέσω και θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Πρώτα απ' όλα το θέμα των υποδομών. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο το ζήτημα. Ο πρόεδρος Επιτροπής εξήγηλε στην πρώτη του ομιλία για ότι η βασική προτεραιότητα είναι τα ομόλογα έργων και αυτά θα τονίσουν την οικονομία της Ευρώπης, οπότε θα ήθελα ε, να τοποθετηθείτε κι εσείς ε, για αυτά τα project bonds, ε, τα ομόλογα έργων επίτροπε, για να δούμε πώς μπορούμε να τα αξιολογήσουμε και νωρίτερα, πριν το 2014. Δεύτερον, τα τεστ κοπόσεως ε, που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά τα τελευταία γεγονότα της ε, Φουκουσίμα γιατί αναβαθμίστηκε στην κλίμακα και έχει φτάσει στο επίπεδο του Τσερνόμπιλ το ατύχημα της Φουκουσίμα οπότε ε, καταλαβαίνετε πόση σημασία έχουν τα ζητήματα πυρηνικής ασφάλειας. Θα είναι ε, υποχρεωτική αυτή η έλεγχη, θα υπάρχουν αμερόληπτες αρχές ε, αξιολόγησης για τα τεστ κόπωσης ε, και τρίτον θα ε, καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα, δηλαδή ε, θα μπορεί να αποφασιστεί το προσωρινό ή το ολοκληρωτικό, ο προσωρινός ή ολοκληρωτικός παροπλισμός των πυρηνικών μονάδων, αν αποτύχει ε, κάποια τέτοια μονάδα το τεστ κοπόσεως. Πρέπει να αντλήσουμε πάρα πολλά διδάγματα από αυτά που συνέβησαν στην Ιαπωνία πέρα από τα τεστ εκοπόσεως. Εμείς ε, θα ε, υποστούμε τεστ υπομονής μέχρι να βρούμε τη λύση. Η πανάκια δεν υπάρχει, θαυματουργή λύση δεν υπάρχει και είναι θέμα ασφάλειας για τους πολίτες. Πρέπει να διδαχθούμε από αυτή την εμπειρία. Ε, τρίτον, ενεργειακή αποδόση συγχαρητήρια γιατί θέτεται και δεσμευτικούς στόχους από το 2014 και μετά για τα δημόσια κτίρια. Αλλά ε, πολύ σωστά είπε μόλις η συνάδελφος Τικάου ότι ναι μεν, ωραία, καλή ενεργειακή απόδοση των δημοσίων κτίριων ε, αλλά μήπως θα έπρεπε να φροντίσουμε και να εφαρμόζεται στην πράξη και το σχετικό νομοσχέδιο. Κάτω των δύο λεπτών σας παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος, δεν προλαβαίνουμε. Ε, η κυρία ε, Τόιερ, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω πολλές σύντομες ερωτήσεις. Πρώτη, εσωτερική αγορά. Πιστεύω πως η εσωτερική αγορά ενέργειας δεν είναι ούτε διάφανες, ούτε προσβάσιμο, ούτε ανοιχτό. Και να σκεφτούμε ότι το δεύτερο ενεργειακό πακέτο υπάρχουν 40 ανοιχτές παραβάσεις. Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει για να ανοίξει αυτή η αγορά, όχι μόνο ε, ανάμεσα στις ε, χώρες ε, πρώην πρωταλτές, αλλά και στο πλαίσιο των νέων χωρών ε, ε, ενεργειακή απόδοση. Είπατε για να υπάρξουν δεσμευτικοί στόχοι εάν δεν γίνει πρόοδος πέραν των δημόσιων τομέα ή άλλοι τομείς βιομηχανική που θα πρέπει να είναι αποδοτική στο τομέα της ενέργειας δεν ε, κάνουν βήματα προς τα εμπρός από ό,τι άγνωστα. Και εδώ θα πρέπει να ποσοτικοποιήσουμε ανακλάδο κάποιες ε, δεσμεύσεις και κάποιους στόχους δημιουργικούς. Το Κοινοβούλιο είχε εγκρίνει με μικρή πλειοψηφία μια, μια απόφαση προς την κατεύθυνση αυτή και είχε συμπεριλάβει την ε, λόγο προβληματική τέλος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν για τις χώρες του Μεσογείου μπορεί να υπάρξει μια μελλοντική ανάπτυξη και βλέποντας, έχοντας τον, το μυαλό μας στο μέλλον, να δούμε όχι τι υπάρχει μόνο στο υπέδαφος, αλλά και τι βρίσκεται πάνω στο έδαφος και να οργανώσουμε κάποιο πρόγραμμα ανάπτυξης και συνεργασίας με τις χώρες αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω μια πολύ σύντομη ερώτηση έτσι ώστε όλοι οι συνάδελφοι να έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν. Ε, έκλεισε το μικρόφωνο του μιλητή. Η στρατηγική και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον τομέα που μας απασχολεί είναι ζητήματα πολύ σημαντικά. Έχουμε κάποιες προθεσμίες, π.χ. το 2020. Θεωρείται ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσουν να θέσουν στην υπηρεσία του ενεργειακού τομέα τα απαραίτητα κονδύλια, κονδύλια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλπ. Ευχαριστώ. Κύριος Διάντζελης. Με ευχαριστώ εντάχει. Μετά από την Φουκουσίμα θα πρέπει όλοι να προβληματιστούμε ειδικά επί της ενεργικής πολιτικής και άρα επί των στρατηγικών που θα ακολουθήσουμε. Εντάξει, σωστά το θέμα της εξωτερικής ενεργικής πολιτικής, αλλά ας μπούμε στην ουσία. Ε, δεν θεωρείται Επίτροπε, ότι έφτασε η στιγμή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, όχι σε ένα, ένα μακρό χρονικό διάστημα, να ε, βελτιώσουμε, να εξυψώσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, να στοχεύσουμε στην καθαρή, στις καθαρές μορφές ενέργειας και ειδικά στις ε, ασφαλείς μορφές ενέργειας. Δεύτερη ερώτηση. Τώρα από πλευράς αυτονομίας και ανεξαρτησίας σε ποιους φορείς θα ανατεθεί η εφαρμογή των stress test ειδικά για να φέρουμε στις καταστάσεις που δεν θα περάσουν αυτό την δοκιμασία το αντοχής και θα πρέπει να ενημερωθεί όπως καταλαβαίνετε η Κομισιόν για αυτές τις δοκιμές. Ευχαριστώ, ο Οντί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω κάτι σχετικά με τα δοκιμές αντοχής. Θα πρέπει να βασιστείτε και να στηριχθείτε στις εθνικές εξειδικευμένες αρχές που έχουν τα υψηλότερα επίπεδα παγκοσμίω. Δεν νομίζω ότι η Κομισιόν έχει την εμπειρία και την ανεξαρτησία για να κρίνει αυτές τις δοκιμές. Ε, τώρα να σας πω κάτι για τις υποδομές, ε, διότι έχουμε μια έκθεση η οποία βρίσκεται στα σκαριά και θα υπάρξει ακρόαση δεν πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει ένας ε, ευρωπαϊκός προβληματισμός αναφορικά με το θέμα της ιδιοκτησίας, ανάπτυξης, εξέλιξης ε, ε, των νεφριών δικτύων και να υπάρξουν καινοτόμες χρηματοδοτήσει που θα στηρίζονται στην κατανάλωση προκειμένου να υπάρξει αλληλεγγύη από όλους τους καταναλωτές όπου και αν αυτοί βρίσκονται στην επικράτηση της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι καταρτίζεται τον οδικό χάρτη μέχρι το 2050. Ποια είναι τα σενάρια μείωσης ε, των ε, αερίων θερμοκηπίου. συμπεριλαμβάνονται στον ε, οδικό αυτό χάρτη. Εγώ έλαβα πολλές τροπολογίες στην έκθεσή μου η οποία αναφέρει μια μείωση του δεξιού του άνθρακο αν του 20% και μια ε, εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και αυτή άνω του 20% μέχρι το 2020. Μέχρι το 2020 πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε αυτούς τους στόχους το 2020. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο τομείς ερωτήσεων. Το πρώτο αφορά τεστ κοπόσεως. Θα λάβει υπόψη η Κομισιόν τα αποτελέσματα των γερμανικών αρχών, ειδικά όσον αφορά την προστασία από πτώσεις αεροσκαφών ή μεγάλες πλημμύρες. Δεύτερον, η Κομισιόν θα προχωρήσει, θα ζητήσει το μορατόριο κατασκευής νέων σταθμών όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το οποίο σας πενθυμίζω ήταν και συμβαστική μα λύση. Και τρίτον, τι άποψη έχει ο Επίτροπος Ενέργειας για τη νέα φορολογία διοξιδίου του άνθρακα που θα αποφασιστεί αύριο στην Κομισιόν. Κάρενς. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Ασφάλεια Πυρηνικών Εργοστασίων. Είπατε πως συζητάτε με τους Ρώσους και Λευκορώσους γείτονες. Το ερώτημα είναι πως θα καταφέρετε να επιβάλλετε τις υψηλές ευρωπαϊκές προδιαγραφές στους γείτονές μας αυτούς. Κυρία Χέρτσογκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο που έρχεται συχνά στην Επιτροπή μας. Βέβαια, εμείς τα, τα δυσκολεύουμε τα πράγματα πολύ, αλλά παρόλα αυτά είναι αναζωογονητική εμπειρία και για τους μεν και για τους δε. Λοιπόν, το πρώτο θέμα. Επί Πολυνικής Προεδρίας θα αρχίσουμε να συμφωνούμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το νέο πλαίσιο. Πώς θα προετοιμαστείτε ούτως ώστε ε, στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου να μεγιστοποιήσετε το δυναμικό που υπάρχει για τα ενεργειακά ζητήματα και πώς μπορούμε εμείς να σας συνδράμουμε. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη είναι και πιο εύκολη. Πόσο ξέρουμε μέχρι το τέλος του ενεστώτος έτους ε, το Αζερμπαϊτζάν τελικά θα αποφασίσει για το πρόγραμμα Ναμπούκο και άλλα συναφή προγράμματα θα αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία. Οπότε, ε, πιστεύετε, ποιο πρόγραμμα πιστεύετε ότι είναι καλύτερο για την Ευρώπη και θα αποφασιστεί μέχρι το τέλος του έτους. Τρίτη ερώτηση που σχετίζεται με τα πυρηνικά ζητήματα. Η οδηγία για την ε, πυρηνική ασφάλεια έχει εγκριθεί, αλλά μόνο έχει, μεταφερθεί στην Εθνική Νομοθεσία τριών μόνο χωρών. Οπότε 24 κράτη-μέλη, εκ των οποίων και ένα που άμεσα εμπλέκεται στα πυρηνικά ζητήματα, δεν έχει μεταφέρει στην Εθνική Νομοθεσία το, την οδηγία. Τι θα κάνετε ε, για να μεταφερθεί πριν αρχίσουμε να τροποποιούμε την οδηγία, γιατί κατά πάσα πιθανότητα μετά τα τεστ κοπόσεω ε, θα κληθούμε να την αναθεωρήσουμε. Και μια προσωπική, ένα προσωπικό σχόλιο. Υπάρχουν ε, κάποιε χώρε που θέλουν να χρησιμοποιούν ένα μόνο κομματάκι του ενεργειακού μείγματο ε, στη δική του επικράτεια. Δεν θέλουν ε, να εισάγουν, δεν θέλουν ούτε να παράγουν πυρηνική ενέργεια, ούτε να εισάγουν πυρηνική ενέργεια. Αλλά εγώ αναφέρομαι στι χώρε που δεν θέλουν να την παράγουν, θέλουν να την εισάγουν. Πώ θα γίνει να το εμποδίσουμε αυτό. Σα ευχαριστώ. Τώρα ο κύριο Επίτροπο έχει τη δυνατότητα να απαντήσει σε ερωτήσει 20 ε, συναδέλφων. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, πρώτα απ' όλα για την οδηγία περί πυρηνικής ασφάλειας, αυτή την εγκρίνατε εσείς τον Ιούνιο του 2009 και θα πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι τον Ιούλιο φέτος. Οπότε τα κρατημέλη που δεν το έκαναν έχουν ε, τρεις μήνες ακόμα περίπου. Και τον Ιούλιο, εκεί όπου δεν έχει εφαρμοστεί η οδηγία, αμέσως μετά θα λάβουμε τα μέτρα μας. Γιατί ειδικά σε αυτό το τομέα δεν είναι δυνατόν να έχουμε καθυστερήσεις και μη εφαρμογή. Το ίδιο ισχύει για την οδηγία πυρηνικών αποβλήτων που ε, εξακολουθεί ε, να είναι στο Συμβούλιο και αναμένουμε από το Συμβούλιο συμπληρώσεις, ε, βελτιώσεις κτλ. αλλά και έγκριση. Γιατί το δίδαγμα που πρέπει να βγει από τη Φουκουσίμα είναι εξαντλημένα καύσιμα δεν μπορεί να παραμένουν γύρω-γύρω από τα πυρηνικά εργοστάσια. Εκεί ε, αυξάνουν τον κίνδυνο. Πρέπει να είναι σε ασφαλείς προσβάσιμες εγκαταστάσεις, υποέλεγχο και προς τα εκεί εργάζεται η οδηγία ε, πυρνικών αποβλήτων. Ήτερ, συνεχίζουμε την έρευνα και θέλω να σας πω ρήτος πως στόχος μου είναι τα μέσα του Ήτερ να μην επιδεινώσουν την χρηματοδότηση των υπολείπων. Έχουμε δηλαδή το ΙΤΕΡ και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Έρευνα που δεν θα πρέπει να υποστεί περικοπές λόγω ΙΤΕΡ επίσης. Καταλαβαίνω πως υπάρχουν θεμελιώδη ζητήματα προϋπολογισμού πλέον όσον αφορά το ΙΤΑΡ, όμως δεν μπορώ να έχω αυτή την ομοιρία κάθε φορά που με ρωτάνε οι Αμερικάνοι και οι Κινέζοι τελικά το θέλετε αυτό το έργο στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει λοιπόν Κοινοβούλιο, Συμβούλιο Κομισιών, να καταλήξουμε σύντομα σε κάποιο αποτέλεσμα, το συντομότερο δυνατόν. Όσον αφορά τα τεστ κοπόσεω, δεν είναι πανάκια. Αλλά, σας λέω ξεκάθαρα, ε, καλύτερο να γίνουν παρά να μην γίνουν. Γιατί βεβαίω. χωρίς αυτά τα τεστ έχουμε ε, λιγότερα στοιχεία στη διάθεσή μας και λιγότερη πειθό. Οπότε επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή τα κριτήρια εξέτασης και μέσα Μαΐου θα συναντηθούμε τις εθνικές εποπτικές αρχές και θα μιλήσουμε για μια πρώτη πρόταση των ε, κριτηρίων. Θα πρέπει να έχουμε πλήρη διαφάνεια γιατί η αυθεντία, η εγκυρότητα των τεστ αυτών εξαρτάται ακριβώς από τη διαφάνεια για να μπορεί κανείς να απορρίψει εύκολα τα αποτελέσματά τους. Μιλάμε επίσης για υψηλότατες προδιαγραφές ασφαλείας. Αλλά, ξέρετε, τι εννοούμε υψηλότατες. Ε, αυτό είναι σχετικό στον καθένα. Δηλαδή όταν μιλάμε για σεισμούς και κίνδυνο από σεισμούς οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε εκεί πολύ ψηλές προδιαγραφές. Πλημμύρες επίσης. Ε, θέμα κυρίως μας αποσχολεί στον Ατλαντικό, όχι στα εσωτερικά ύδατα. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει ενίσχυση με τα απαραίτητα μέσα όπου είναι δυνατόν. Επίσης, συστήματα ψήξης και η λειτουργία τους. Γεννήτριες ανάγκης και η διασφαλισμένη λειτουργία τους. Πράγματα τα οποία νομίζω μπορούν να λυθούν με συνένεση. Τώρα, πτώσεις αεροσκαφών, ανεξαρτήτως του εάν είναι επίθεση ή ατύχημα. Τι ξέρω εάν θα έχουμε το υψηλότερο επίπεδο σε όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί σαφές είναι πως εάν έχουμε μία επίθεση όπως στο Σεπτέμβριο του 2001 στη Νέα Υόρκη, δηλαδή μια εσκεμμένη τρομοκρατική ενέργεια, ε, τότε κανένα πυρηνικό εργοστάσιο στον κόσμο δεν είναι επαρκώς εξασφαλισμένο και ίσως να μην είναι και τεχνικώ δυνατόν ή δεν ε, συμφέρει οικονομικά. Οπότε πρέπει να αποφασίσουμε εάν ε, θα δεχτούμε ένα βαθμό κινδύνου. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να δούμε και το εάν το δέχεται αυτό ένα κράτος μέλος, γιατί βεβαίω, όπως ξέρετε έχει την δυνατότητα να αποφασίσει το ενεργειακό του μείγμα, γιατί ξέρετε πως έχει πολλές ε, δυνατότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν μπορεί να πει ποιο θα είναι το ενεργειακό μείγμα μιας χώρας. Ξέρετε πως η Γαλλία και η Αυστρία είναι 38 παραδείγματα. Τώρα, για αυτό το οποίο είπατε κύριε Χέρτσογκ, θα γίνει και στη χώρα μου. Ξέρετε, προτάθηκε απαγόρευση εισαγωγής ε, ε, ρεύματος από πυρηνικής ενέργειας. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει γερμανικό και λουξεμβούργικο ρεύμα. Υπάρχει ρεύμα στην εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά δεν διακινείται επαρκώς διασυνοριακά, αλλά υπάρχει μια κοινή βούληση να υλοποιήσουμε την εσωτερική αγορά και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς. Αλλιώς δεν θα γίνεται τίποτα. Δηλαδή πηγαίνει από την ε, Ισπανία στη Γαλλία, από τη Γαλλία στη Γερμανία, από την Γερμανία στην Τσεχία Έχουμε δηλαδή μια ευρωπαϊκή αγορά και θα πρέπει να έχουμε μακροπρόθεσμες συμβάσεις και αυτό σημαίνει πως όποιος θέλει να απαγορεύσει το ρεύμα από πυρηνική ενέργεια ή από άνθρακα ή αντιστρόφως από αιωλική ενέργεια δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και ξέρετε, ε, δίνουμε λεφτά ε, στη γεωργία για απόσταση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και διάφορα πράγματα, θα πρέπει να ε, δώσουμε λεφτά και για την ενέργεια. Τώρα, για τις εξαγωγές. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε επίσης τις εξαγωγές Τώρα, όσον αφορά χώρες γειτονικές και την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, όταν μιλάμε για τη Ρωσία παραδείγματο χάρη και το Καλίνιγκραντ. Κοιτάξτε, θέλουν και οι Ρώσοι να μας πουλήσουν ρεύμα από το Καλίνιγκραντ. Όχι μόνο φυσικό αέριο και πετρέλαιο και άνθρακα, αλλά και ρεύμα. Και εμείς θέλουμε να πουλήσουμε αυτοκίνητα στη Ρωσία. Οπότε τι θα κάνουμε. Εάν αμυνθούμε και πούμε δεν θα έχουμε εισαγωγές ε, ρεύματος, τι θα κάνουμε, θα πούμε όχι ή θα πούμε πως το αποδεχόμαστε αλλά πρέπει να έχουμε προδιαγραφές ασφαλείας. Και βεβαίω αυτό το θέμα αφορά όλη την αγορά ρεύματο Πολωνία και Βαλτικών χωρών. Τώρα για τον Τέζερτεκ. Περί τίνο πρόκειται. Κοιτάξτε. Εμφύλοι πόλεμοι ή ε, μη εμφύλοι πόλεμοι. Πρέπει να υπάρχει μια εταιρική σχέση με τη Μεσόγειο και όχι μόνο club med και διακοπές. Θα πρέπει. Να δούμε. Και ε, δύο πράγματα. Το ένα αφορά βεβαίως ε, τη γεωργία και τα γεωργικά προϊόντα και τους αγρότες, ε, τους Ευρωπαίους, Ισπανία, τα κτλ. Και το δεύτερο βεβαίως την ενέργεια. Ξέρετε, οι πετρελαιοπαραγωγές χώρε καίνε πετρέλαιο για να παράξουν ρεύμα. Εμείς δεν το κάνουμε πλέον, δεν είναι η τελευταία τεχνολογία εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε, τι θα ήταν ιδεώδες για το κλίμα μας. Άμεσα ενέργεια από τον ε, ήλιο και αργότερα κύματα και αέρας και να διηγηθούμε από εκεί και στην κινητικότητα κτλ. Αλλά βεβαίως εκεί πέρα με το πετρέλαιο έχουν μία κιλοβατόρα με 2,5 σέντ ενώ με την ηλιακή ενέργεια χρειάζονται 6 σέντ. Οπότε ένα μεγάλο ποσοστό θα πρέπει να καλυφθεί από επιδοτήσεις. Αλλά αυτό σημαίνει να γίνουν ενιαίοι οι κανονισμοί οι ευρωπαϊκοί των ε, ανανεώσιμων πηγών. Και αυτό είναι ευαίσθητο. Ξέρετε και στη Γερμανία. Γιατί. Αν έχουμε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις εκεί πέρα που, χρειάζονται, που θα μπορούσαν να έχουν 2.500 ώρες ηλιοφάνεια το χρόνο, έχουν μόνο 800. Αλλά ξέρετε, από μόνοι τους ε, Αλγερινοί και Λίδοι δεν θα κάνουν κάτι τέτοιο, γιατί έχουν αρκετό πετρέλαιο και μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό. Οπότε το θέμα είναι πώς θα οργανώσουμε μια επιδότηση, μειωμένη επιδότηση, που βεβαίως θα έχει πολλαπλό αποτέλεσμα για το διοξείδιο του άνθρακα. και θα είναι πιο αποτελεσματικό από μέτρα ακριβότερα εντός της Ευρώπης. Και άρα δίνουμε βάση σε αυτό για την μείωση αυτή του 20% να μην είναι μόνο εντός της Ευρώπης αλλά και με ευρωπαϊκά μέτρα εκτός της Ευρώπης. Γιατί το κλίμα δεν είναι ευρωπαϊκή υπόθεση, είναι παγκόσμια. Και προετοιμάζουμε τις, την επόμενη βεβαίως δημοσιονομική περίοδο η πρόταση της Κομισιόν θα έρθει τον Ιούλιο και είμαι σίγουρος πως για την ενεργειακή έρευνα θα έχουμε επαρκή μέσα. Δεύτερον, για την ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Θεωρώ πως η συνοχή των διαρθρωτικών προγραμμάτων είναι σωστά γιατί μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με λίγη γραφειοκρατία και είναι σωστό ούτως ή Και η προτεραιότητα στην Κομισιόν και στα κράτη-μέλη ε, είναι κοινή. Τρίτον, υποδομές διασυνδέσεις, ε, δίκτυα κτλ. Εκεί θα κάνουμε την πρόταση ομολόγων έργων υποδομών για πληροφορική, συγκοινωνίες και ενέργεια. Ή και ενέργεια μόνα τους. Και το συναπαστικό ερώτημα θα είναι το εάν τα κράτη-μέλη θα αποδεχτούν τα ε, ομόλογα. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ε, λαμβάνονται αποφάσεις για προτάσεις που γίνονται. Είτε μιλάμε για φορολογία, ενέργειες, είτε για φόρο ε, χρηματοοικονομικών ε, συναλλαγών. Και π.χ. στη δική μου χώρα, από την κυβέρνηση την, του δικού μου κόμματος, μια κυβέρνηση συνασπισμού βεβαίω συμφώνησε να πει πως ευρωπαϊκός φόρος τέτοιος δεν θα υπάρχει. Και ευρωπαϊκός φόρος κανένας δεν θα υπάρχει. Δεν είναι πολύ φιλικό προς την Ευρώπη γιατί θα πρέπει τα κράτη-μέλη τουλάχιστον όσον αφορά τα ομόλογα αυτή την ε, εγγύηση για να δημιουργηθούν υποδομές να την δεχτούν τουλάχιστον. Μετά ακούστηκε το ερώτημα το πώ θα προωθήσουν περισσότερο τι ανανεώσιμε πηγέ. Κυρίε και κύριοι, είμαστε σε επιτυχή ε, δρόμο. Γιατί το 20% μέχρι το 2020 είναι μέρος τη εικόνας. Γιατί αν δείτε τις μεταφορές θα έχουμε επιτύχει μόνο το 10%. Γιατί δεν θα υπάρξει π.χ. αλλαγή στα αεροπλάνα, στα φορτηγά κτλ. Και όταν φτάσουμε στα Αγιώταχη, μιλάμε για καμιά δεκαετία που θα έχουμε φτάσει ένα 10% το πολύ μιλάμε. Αλλά στον τομέα της παραγωγής ρεύματος. Θα πρέπει άρα να φτάσουμε στο 35% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε θα ξεπεράσουν το 2014-2015 ε, ήδη τον άνθρακα. Αλλά ξέρετε πως αυτό δεν μπορεί να γίνει δεσμευτικό να πάμε παραπέρα από το 20% γιατί δεν το δέχονται κάποια κρατημέλη. Αλλά χρειαζόμαστε άρα και μια προοπτική παραπέρα. Γιατί το θέμα τι θα γίνει περαιτέρω είναι ένα σημαντικό ερώτημα το οποίο πρέπει να δούμε τώρα. Βεβαίω κύριε Γκέμπελ, έχετε δίκιο. Ε, δεν ξέρουμε ποιε θα είναι οι τεχνολογικέ εξελίξεις. Αλλά όταν μιλάμε π.χ. για το 2050 το ότι η παραγωγή ενέργειας δεν θα πρέπει να εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα είναι κάτι το τεχνικά εφικτό ως μακροπρόθεσμη στρατηγική. Και άρα είναι απόφαση του, Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να πούμε πως το 2050% να έχουμε 80% λιγότερες εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα. Και άρα έχουμε πρώτον ανανεώσιμες, δεύτερον δέσμευση και αποδίκευση στα άνθρακα και τρίτον, εάν δεν αλλάξει τίποτα στα κράτη-μέλη, και πυρηνική ενέργεια. Και κύριε Μπιουτικόφερ, θα έχουμε και ένα σενάριο με αντικειμενικά δεδομένα, κόστος και λοιπά, με 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα 40 χρόνια μέχρι το 2050. Haben beim Binnenmarkt Έχουμε μια εσωτερική αγορά λοιπόν Έχουμε λοιπόν το τρίτο πακέτο της εσωτερικής αγοράς που πρέπει να εφαρμοστεί από το Μαρτίο πρέπει να έχει εφαρμοστεί. Λέμε στα κράτη-μέλη τι δεν έχουν κάνει, ε, που δεν έχουν κάνει αρκετά πράγματα. Διαβουλευόμαστε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν δύσκολα νομικά θέματα και αντιδράσεις και ε, τουλάχιστον το αργότερο το φθινόπωρο θα ξεκινήσουμε διαδικασίες σε παραβάση. Γιατί βεβαίως όπως σας είπα και η αποδέσμευση είναι σημαντικό σημείο, σημείο κλειδί εδώ πέρα. Και κοιτάξτε τι θα χρειαζόμασταν. Θα χρειαζόμασταν μια αστυνομία εσωτερικής αγοράς. Αν πάμε σε ένα κράτος μέλος και βλέπουμε διαπλοκή κράτους και επιχειρήσεων ενέργειας. δεν υπάρχει διαφάνεια και βλέπετε πως είναι για κάποιους κυβερνώντες πολύ σημαντικό μέσο. Και μιλάμε για πολύ μεγάλα κράτη-μέλη. Οπότε, εγώ χαίρομαι για το ότι το 2014 θα έχουμε ολοκληρώσει την εσωτερική αγορά της ενέργειας. Είναι φοβερή πρόκληση. Και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τα επόμενα δύο χρόνια θα απορούν και πώς θα πρέπει να εφαρμόσουν τις ίδιες τους τις αποφάσεις. Όπως σας είπα, έχουμε κάνει, δεν ξέρω, ένα 40% ε, των όσων θα έπρεπε να έχουμε κάνει. Ενώ ξέρετε, σε πάρα πολλά άλλα ήδη υπάρχει ουσιαστικά η εσωτερική αγορά. Ε, τώρα, όσον αφορά τα ιδιωτικά ακίνητα, θα πρέπει βεβαίως και αυτά να ενταχθούν στο πρόγραμμά μας όσον αφορά την κατασκευή νέων κατοικιών. Πράγματι μπορεί να υπάρξει ενίσχυση για την ανακαίνιση τους και βεβαίως και συγκριματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος σας υπόσχομαι πως η ανακοίνωσή μας για την εξωτερική ενεργειακή πολιτική θα υποβληθεί πρώτα απ' όλα σε εσάς για εμένα εσείς είστε η βασική επιτροπή. Γιατί μιλάμε για ενέργεια πρώτα απ' όλα και σε δεύτερο λόγο για εξωτερική πολιτική. Αλλά βεβαίως μιλάμε για μεγάλες στρατηγικές σχέσεις όπου θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε ποια είναι τα γενικότερα συμφέροντά μας. Δηλαδή μιλάω εδώ πέρα για South και Ναμπούκο ή Ναμπούκο και IDGI. Προσπαθούμε να έχουμε μια συνολική λύση, αλλά δυστυχώς διαπιστώνω πως το roadshow των Ρώσων ε, συνεταίρων μας καταραίει. Οπότε, όταν μιλάμε για ε, για εξωτερική πολιτική ενεργειακή πρέπει πρώτα και εσωτερικά να έχουμε μία συνοχή. Και δεν είναι δυνατό να επιτρέπουμε να εφαρμόζουν οι Ρώσοι το Διέρη και Βασίλευε σε εμάς. Και για το θέμα της ε, φορολόγησης ενέργειας ο κύριος Σεμέτα θα έρθει αύριο στην ε, Επιτροπή γι' αυτό έχω σοβαρές αμφιβολίες επιφυλάξεις Υποθέτω πως η μεταβατική περίοδος θα πάει μέχρι το 2023, αλλά η άποψη στην Κομισιόν είναι να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα τώρα. Ποιο είναι λοιπόν το ζήτημα. Το πετρέλαιο και τα προϊόντα βενζίνη κτλ. να φορολογήσουμε με την, ενέργεια, την περιεκτικότητα σε ενέργεια. Δηλαδή να μην φορολογούμε το λίτρο, αλλά την ενέργεια που περιέχει, που περιέχεται περισσότερη σε ένα λίτρο ντίζελ. Οπότε λένε πως η ελάχιστη φορολογία στο λίτρο με, ε, που είναι γύρω στο 40 cent δεν είναι πρόβλημα και ξέρετε σε πολλές χώρες είναι υψηλότερη αλλά εάν φορολογήσουμε με βάση την ενέργεια που περιέχεται τότε θα πρέπει ε, το ντίζελ να φορολογηθεί κατά 17% παραπάνω και είτε θα μειωθεί η βενζίνη είτε θα αυξηθεί το ντίζελ. Έχω αμφιβολίες για τον εξή λόγο. Κοιτάξτε, έχουμε άλλα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Ε, δεν ανάγκη να δίνουμε και θέματα στον κίτρινο τύπο, αλλά όπως είπα η Κομισιόν αποφασίζει συλλογικά και θεωρεί πως πρέπει να, να το κάνουμε αυτό και κοιτάξτε, ούτω ή άλλω ε, είναι θέμα των, των κρατών μελών. Το τι θα γίνει με αυτήν την ομορφή. Σα ευχαριστώ γιατί ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση κύριε Επίτροπε. Γιατί ε, είχαμε συγκεκριμένε ερωτήσει και απαντήσει. Και αυτό βεβαίω βοηθάει. Γιατί δεν έχουμε μόνο λόγους, αλλά ε, και αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, κύριε Επιτροπέ. Darf dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur nächsten, zum nächsten... Περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερησίας διάταξη. ενεργειακή υποδομές, προτεραιότητες μέχρι το 2020 και παραπέρα. Συνάδελφοι, θέλουμε να δούμε και τα υπόλοιπα σημεία της ημερήσιας διάταξης και οι συνάδελφοι που είναι αρμόδιοι θέλουν και αυτοί να ακουστούν και να μιλήσουν. Μήπως λοιπόν οι συζητήσεις ε, που δεν αφορούν αυτό το θέμα να περάσουν έξω και να δώσουμε τον λόγο μόνο στον Σόζο Βάγνερ που είναι ο εισηγητής μας και ε, είναι ο μόνος που έχει τον λόγο. Σας παρακαλώ κύριε και κύριοι. Ο εισηγητής έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος ε, και τα μέλη συνάδελφοι αυτής της Επιτροπής ε, καταλαβαίνουν πως όταν είδα τις 600 περίπου τροπολογίες ε, που μου έπεσαν στο κεφάλι θεώρησα πως ε, πρόκειτο για ένα μαρτύριο παρόμοιο με αυτό που αναφέρει ο Δάντες Αλιγέρης ε, στην ε, Θεία Κομωδία και δει στον, στην κόλαση. Αλλά διαβάζοντας όμως τις ε, διάφορε τροπολογίες κατα... κατάλαβα πως η Θεία Πρόνοια ήταν, φέρθηκε ιδιαίτερα ευνοϊκά διότι οι τροπολογίες που ενώ στην αρχή θεώρησα ότι πρόκειται για ένα θείο μαρτύριο αφορούσαν ε, στην ε, περαιτέρω βελτίωση και αποσαφήνιση του κειμένου και ως εκ τούτου να το εμπλουτίσουν. Θεωρώ λοιπόν πως θα είναι σχετικά απλό και εύκολο να δουλέψουμε επί των τροπολογιών προκειμένου να καταλήξουμε σε συμβασμούς και σε διάφορους κανόνες που θα μας ε, ικανοποιούν όλους. Τώρα, ε, εγώ ως και σε συνεργασία με τους βοηθούς αλλά και με τους ε, σκιώδη ηγητέ θα συνεργαστούμε. Θεώρησα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσε τι τροπολογίε ε, που κατατέθηκαν και που τόνισαν την σημασία της εσωτερικής αγοράς ενέργεια και της ε, ασφάλειας ε, αυτών των δικτύων. Αυτό προέκυψε από τη συζήτηση που είχαμε μέχρι τώρα, τη συζήτηση που είχαμε και με τον αρμόδιο επίτροπο, αλλά θα ήθελα να τονίσω το ζήτημα και να πω ότι στην Ήπειρό μας, στην Ευρώπη μας ε, έχουμε κάποια προβλήματα επισφάλειας ε, στον τομέα της ενέργειας, είμαστε ευαίτερα ευάλωτοι και υπάρχουν πολλές χώρες που εξαρτώνται από έναν και μόνο προμηθευτή. Είναι χώρες ε, που θα λέγαμε ότι είναι όμοιροι. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να αλλάξουμε την κατάσταση, να ενεργοποιηθούμε μια που μιλάμε για ενέργεια. Τώρα θα ήθελα να πω πως ε, σημαντική είναι η άποψη σύμφωνα με την οποία ε, η ζήτηση της ενέργειας θα πρέπει να συνδεθεί με τις ε, υποδομές οι οποίες πρέπει να τύχουν κάποιες ιεράρχησης δεν νομίζω ότι θα πρέπει να δρούμε με τρόπο ε, ακατάστατο δημιουργώντας ενεργικές υποδομές ε, ή, ή ενεργικές διασυνδέσεις ε, θεωρώντας ότι από μόνο του αυτό είναι κάτι το θετικό, κάτι το καλό. Θα πρέπει να έχουμε αναλύσει τις όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν, την ζήτηση που υπάρχει στον τομέα της ενέργειας και την ε, ενεργειακή απόδοση. Να δούμε λοιπόν ποια είναι τα στοιχεία κλειδιά που θα μας βοηθήσουν για να προσδιορίσουμε τις ανάγκες μας. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ανταποκριθούμε με τις ε, ικανές υποδομές λίγος να υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις. Αυτό αναφέρεται στην έκθεση, αλλά Θεωρώ πως οι τοπολογίες που έχουν κατατεθεί ε, τονίζουν αυτά τα οποία εγώ έχω γράψει στην εκθεσία μου. Επίσης, ε, ιδιαίτερη προσοχή αποδίδω στα κριτήρια προκειμένου να επιλέξουμε. Μπορούμε να μιλήσουμε για απαιτήσει ε, που θα πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια για, την, για να επιλεγούν αυτές οι υποδομές. Συζητήθηκε το ζήτημα αυτό στις συζητήση που είχαμε μέχρι τώρα, ποια θα είναι τα κριτήρια μέσω των οποίων θα επιλέγουμε, να λέμε ότι αυτό ενδιαφέρει και είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης, αυτό δεν έχει, την χάνει προτεραιότητας, ε, αυτό όχι. Ε, Παντώντα λοιπόν σε αυτές τις ερωτήσεις, ε, θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μια αποτελεσματική πολιτική ε, υποδομών ενέργειας. Οι τροπολογίες λοιπόν αναμφίβολα συμβάλλουν στο να διευκρινίσουν ότι τα σημεία 24 και 25 της εκθέσεώς μου ε, είναι σημεία τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε κάποια σύγχυση. Χρειάζεται λοιπόν να ξεκινήσουμε από τους στόχους της ενεργικής πολιτικής αφενός, στόχους που για μας έχουν καταστεί σαφείς διότι εμείς βασιζόμαστε στους στόχους που περιέχονται στις ε, συνθήκες ε, και ξεκινώντας από αυτούς τους στόχους θα πρέπει να καθορίσουμε τις προϋποθέσεις ώστε οι υποδομές να μπορέσουν να αξιοποιηθούν κατάλληλα. Οι προτάσεις λοιπόν που γίνονται θα πρέπει να είναι συνεπείς με την κλιματική πολιτική, με την περιβαλλοντική πολιτική, με τα δίκτυα διανομής που σχεδιάζονται και με άλλες ε, βασικές επιλογές ε, ε, γενικότερης πολιτικής ή βιομηχανικής πολιτικής. Αυτά, αυτή λοιπόν θα πρέπει να είναι οι προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα. Τώρα, έχουμε επίσης και τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο σημείο 25 της εκθέσεώς μου. Αυτά τα κριτήρια θα χρησιμεύσουν για να μπορέσουμε να κάνουμε την κατάλληλη επιλογή των, των προγραμμάτων τερματισμός της ύπαρξης ενεργειακών νήσων, οικονομική απόδοση, καλύτερη σχέση ανάμεσα στο κόστος και την ωφέλεια, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, περιορισμός της συρρήκνωσης των πιθανών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όλα αυτά είναι σημεία τα οποία συμπεριλαμβάνονταν ήδη στην εκθεσή μου, αλλά μετά από τις τροπολογίες που κράτησαν στην άλφη τονίζονται περαιτέρω και απαιτούν ε, μεγαλύτερη ουσία, περισσότερη ουσία. Και είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία με τους συντάκτες των τροπολογιών, ε, Ό,τι αφορά τώρα τις διαδικασίες, ε, τις αδειοδοτήσεις, τις άδειε κλπ που είναι κάτι που μας απασχόλησε αυτής εξ αρχής πιστεύω πως οι τροπολογίες που δεν ζητούν από την Επιτροπή να ε, φτάσει σε μια εναρμόνιση η οποία είναι αμφίβολης ε, ε συνταγματικότητας θα με βάση τις συνθήκες και οι τροπολογίες που αφορούν το να χορηγηθούν στην Κομισιόν αρχές προκειμένου να εποπτεύει τις εθνικές δημόσιες αρχές και άρα τα κράτη-μέλη ε, προκειμένου να πληρούν τους ε, προθεσμίες θεωρώ ότι αυτές οι προθεσμίες δεν ε, τηρούνται εγώ γνωρίζω τι συμβαίνει στην χώρα μου και γνωρίζω πάνω κάτω και το τι συμβαίνει στην Γερμανία. Στην Ισπανία η παράλυση αυτών των ε, προγραμμάτων είναι μια σταθερή. Στην Γερμανία η παραγωγή που γίνεται στη Βόρειο θάλασσα και που προωθείται στην ε, κεντρική Ευρώπη έχει οδηγήσει σε, έχει παράλυση διότι απαιτούνται εκατοντάδες ε, χιλιόμετρα εγκαταστάσεων ε, και ε, υποδομών, υπάρχουν διάφορες προσφυγίες στα δικαστήρια, υπάρχουν διαφωνίες με τις δημόσιες αρχές κλπ. Γι' αυτό χρειάζεται να εξαιρεθεί μια λύση, μια λύση η οποία περνάει όχι από τα εναρμόνιση των εθνικών, ε, των ε, εθνικών δικαίων, αλλά μέσω της ε, δημιουργίας κάποιων μάλλον τη δυνατότητα να χωρίσει στην Κομισιόν κάποιων περισσότερων αρμοδιοτήτων για να μπορεί να ελέγχει τις εξελίξεις. Επίσης θα πρέπει να παροτρύνουμε την ε, πιο συμμετοχική προσέγγιση και να αναγνωρίσουμε πως η διασφάλιση μοναδικής αποδοχής των σχεδίων έργων ενεργειακής υποδομής από τους ε, πληθυσμούς εξαρτάται και από τη συμμετοχή τους ε, σε αυτά τα προγράμματα και στις αποφάσεις. δίχως ε, την στήριξη των ε, κοινωνιών δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Κλείνει το μικρόφωνο του ομιλητή. Πάνω. Τώρα σε ό,τι φορά το τελευταίο κεφάλαιο, η ε, χρηματοδότηση δηλαδή, θεωρώ ότι η εξέβρεση πόρων για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων είναι κάτι το οποίο θίγουν και η εκθεσή μου, αλλά το θίγουν και οι τροπολογίες. Δεν γινόταν αναφορά στην εκθεσή μου πάνω στους, ε, στα δύο ταμεία, αλλά τώρα πιστεύω ότι τα δύο ταμεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη το πνεύμα της πολιτικής συνοχής που διέπει αυτά τα ταμεία. Τώρα δέχομαι επίση τις τροπολογίες ε, που ζητούν να αναφερθούν συγκεκριμένες ε, γεωγραφικές περιοχές όπως ε, η Κομισιόν αναφέρεται σε συγκεκριμένους διαδρόμους αλλά δεν συμφωνώ να δεχθούμε συγκεκριμένα προγράμματα με όνομα και επώνυμο. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, οι εργασίε συνεχίζονται, μπαίνουμε σε μια νέα φάση ε, την εξέταση αυτών των τροπολογιών που είναι μια φάση η οποία θα στηριχθεί σε μια εποφελή και καρποφόρο συνεργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Εφτά ομιλητές θα ακολουθήσουν. Και έχουμε και άλλο ένα σημείο, οπότε κατανότα το άριο 20 λεπτά και όχι παραπάνω. ¿eh? Ε, Κύριε Σόζα Βάγνερ, νομίζω πως ε, εκτός από Θεία πρόνοια με τη δουλειά σας καταφέρατε να συντάξετε μια καλή έκθεση. Σας συγχαίρω λοιπόν για την εργασία σας και θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου ε, αναλύοντας τώρα τις τροπολογίες που, έλαβα, που οι συνάδελφοι από την πολιτική μου ομάδα, διαπίστωσα ένα υψηλό βαθμό σύμπτωσης και συμφωνίας με τα θέσεις του εισηγητή, αλλά επιτρέψτε μου κάποια σύντομα σχόλια. Κοιτάξτε. Τα δύο βασικά θέματα ήταν η χρηματοδότηση μέσω των ομολόγων και την φόρο επί του άνθρακα που νομίζω ότι θα τύχουν της στήριξης του κυρίου Σώσα Φάκνερ θα ήθελα να σχολιάσω πως οι τροπολογίες που έχουν καταθέσει οι σοσιαλιστές συνάδελφοι θα μπορούσαμε να τις ομαδοποιήσουμε σε τρεις ομάδες. Μια πρώτη ομάδα ε, αποτελείται από ένα σύνολο τροπολογιών που ζητούν με ένα μεγαλύτερο επίπεδο ε, ενεργειακή απόδοσης και από ασφαλικότητα ε, και που ζητούν επίσης ε, να διασφαλιστεί η ηλεκτρική κινητικότητα και την ενσωμάτωση των δικτύων Τώρα, μια άλλη ομάδα τροπολογιών τονίζουν την εφαρμογή του τρίτου πακέτου της ιστορικής αγοράς και ένα τρίτο, μια τρίτη ομάδα που αναφέρει την, σαν ανησυχίε για την ε, ανισο, ανισορροπία των μελλοντικών υποδομών σε σχέση με το δημογραφικό πρόβλημα. Αυτές νομίζω ότι είναι τροπολογίες που βελτιώνουν την ήδη πολύ καλή έκθεση του κυρίου Σόζα και όπως είπε ο εισηγητής εύκολα θα μπορέσουμε να καταλήξουμε συμφωνία. So, Karens. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μα σε τρία μόνο σημεία. Ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποιε θα έπρεπε να είναι μάλλον οι προτεραιότητες, πώς να βρούμε την απαιτούμενη χρηματοδότηση για να διαμορφώσουμε την υποδομή που χρειαζόμαστε βάσει των προτεραιοτήτων και τρίτον ε, πώς να καταστήσουμε ευχερέστερη την διαδικασία επιδοτήσεων. Για την παράγραφο 24 έχουμε υποβάλει νομίζω 100 τροπολογίες συνολικά όλοι, αν τις μέτρησα καλά. Πολλές επαναλήψεις βέβαια, αλλάζει η σειρά κτλ. Αλλά φαίνεται να υπάρχει μία ομοθυμία, φαίνεται να ομονώνει οι πολιτικές ομάδες. Δύο ε, βασικές προτεραιότητες ε, φαίνεται να υπάρχουν. Και σας θυμίζω ότι οι προτεραιότητες είναι τα προγράμματα που δύσκολα θα βρουν ιδιωτική χρηματοδότηση ή θα είναι ανέφικτο να βρεθεί ιδιωτική χρηματοδότηση για αυτά. Γιατί για όσα προγράμματα είναι οικονομικά βιώσιμα δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Η αγορά θα μας πει ποιο είναι το πιο σημαντικό. Όμως, όταν μιλάμε για τη δημόσια χρηματοδότηση, νομίζω είναι σημαντικό να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες για να λειτουργήσει εσύ η εσωτερική αγορά θα πρέπει να αποδώσουμε έμφαση σε αυτή στην κατάργηση των ενεργειακών νήσων και την άρση της ε, ενεργειακής εξάρτησης. Νομίζω ότι αυτό προκύπτει από πολυάριθμες τροπολογίες. Επίσης, ε, οι τροπολογίες που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, κοιτάξτε, θα χρειαζόμαστε υποδομή ώστε να πάρουμε από τη Βόρεια Θάλασσα την νεολική ενέργεια και να τη χρησιμοποιήσουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Νομίζω ότι ε, αυτό είναι μια προτεραιότητα και δεν βρίσκει απάντηση μόνο με τα εμπορικά συμφέροντα. Τώρα, πώ θα βρούμε τη χρηματοδότηση. Πρέπει να είναι καινοτόμα. Νομίζω συμφώνησαν όλοι οι συνάδελφοι. Και διαφωνώ με αυτού που είπαν ότι χρειαζόμαστε νέου φόρου για το διεξίδιο του άνθρακα και δεν ξέρω εγώ γιατί για να χρηματοδοτήσουμε τα προγράμματα. Δεν χρειάζεται τρίτον. Χρειάζεται απλουστευμένη και ταχύτερη διαδικασία για την υποβολή προσφορών και ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι και εγώ σύντομη. Θα σχολιάσω κάποια σημεία που, στα οποία πρέπει να ενισχύσουμε κατά τη γνώμη τη θέση του Κοινοβουλίου. Πρώτον, τα κριτήρια επιλογή των προγραμμάτων, ε, το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον έχει καθοριστική σημασία. Ε, κυρία Σόσα Βάγνερ, ελπίζω, ε, ε ο κύριο Σόσα Βάγνερ, ε, ελπίζω να υποβάλει και συμβαστικέ τροπολογίε για τι παραγράφου 24 και 25 για να φανεί ότι χρειάζεται ιεράρχηση προτεραιοτήτων και επίση η ε, να δείξουμε ότι και ο αυξημένος ανταγωνισμός αλλά και η ασφάλεια στον ενεργικό ε, ανεφοδιασμό έχουν ε, την ίδια σημασία, την ίδια βαρύτητα. Στην παράγραφο 7 επίσης πρέπει να τονίσουμε τη σημασία των χρηματοδοτικών μέσων, όπως παραδείγματο χάρη τα ομόλογα έργων, τα project bonds, διότι με πεπισμένη τα κράτη-μέλη ποτέ δεν μπορέσουν να βρουν όλες αυτές τις επενδύσεις για να έχουν τις απαιτούμενες υποδομές χωρίς αυτά τα ομόλογα έργων. Πρέπει να περάσουμε χειρότατο μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτή σαφώς είναι η θέση του Κοινοβουλίου για αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Βιντάλ Κουάντρος τώρα. Ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά Σώσα, δεν πρόκειται για ένα μαρτύριο αυτές οι 600 ε, τροπολογίες. Απλά είναι ένα ε, αφιέρωμα θα έλεγα στον βωμό αυτής της ε, εκθέσεως. Η έκθεσή σας ε, είναι πολύ καλή και οι τροπολογίες θα την βελτιώσουν έτσι περαιτέρω. Είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποιες κατευθύνες γραμμές, στις οποίες όλοι συμφωνούμε και είναι αυτές που θα δώσουν στην έκθεσή σας ε, την ουσία της. Π.χ. η ιδέα που επανειλημμένως αναφέρεται ότι ε, πέρα, εκτός από έναν κατάλογο προγραμμάτων συγκεκριμένων χρειαζόμαστε σωστά κριτήρια και σωστές ε, γενικές αρχές που θα προσανατολίσουν την πολιτική των υποδομών. Αυτό είναι μια ιδέα κλειδί που περιλαμβάνεται σε πολλές τροπολογίες και επί των οποίων φυσικά θα συμφωνήσουμε. Τώρα, η αγορά θα είναι ο βασικός μηχανισμός που θα προωθήσει και θα απαιτήσει τις υποδομές, αλλά πολύ συχνά το διοικητικό άχθος ε, που επιβάλλει η νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο είναι κάτι το οποίο παρεμποδίζει την ε, αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειάζεται αυτό το άχθος να μην είναι υπερβολικό. Το ίδιο συμβαίνει και με τις άδειε και τις ε, αδειοδοτήσεις ε, που καθυστερούν τις διαδικασίες, κάτι το οποίο αποτρέπει ή ονδήποτε επενδυτή ο οποίος είναι διατεθειμένος ε, να χρηματοδοτήσει ένα σχέδιο. Και κάτι ακόμα. Είναι υποχρέωση των κρατών μελών όχι μια εθελούσια συνεισφορά, είναι μια υποχρέωση των κρατών μελών να συνεργαστούν στην οικοδόμηση της εσωτερικής αγοράς ε, των τομέα της ενέργειας. Ως η Κομισιόν που είναι ο ε, θεματοφύλακας ε, των συνθήκων θα πρέπει να προσέξει ότι τα κράτη πληρούν και τηρούν αυτήν την υποχρέωση και να μην εφαρμόζουν διάφορα διοικητικά εμπόδια και να μην δρουν τα κράτη-μέλη σύμφωνα με κάποια πολιτικάντικα κριτήρια και, λαϊ, και ε, λαϊκισμούς. Αυτό ε, είναι κάτι που πρέπει να τηρηθεί και να εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να συγχαρώ λοιπόν τον εισηγητή και είμαι βέβαιο ότι με όλο αυτό το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μα θα οδηγηθούμε σε μια εξαίρετη έκθεση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βάγνερ, περάσατε το στρες το τεστ αντοχής πολύ επιτυχημένα. 600 τροπολογίες και αντέξατε. Η έκθεση είναι εξαιρετική παρότι ήταν μια πολύ δύσκολη έκθεση και δεχτείτε τα συγχαρητήριά μου. κύριε Σιγητά και κύριοι συνάδελφοι, με τον, κύριο, με τον συνάδελφο κύριο Βόμποντα και την κυρία Ποδηματά έχουμε υποβάλει μία παράγραφο στο 28 όπου ζητούμε να γίνουν να γίνει αξιολόγηση των υποδομών, των ενεργειακών υποδομών, αν μπορούν να αντέξουν στις φυσικές καταστροφές. Γιατί βλέπουμε ότι με την αλλαγή του κλίματος έχουμε μέγα φωτιές, ε, μέγα παλιριακά ε, κύματα, μέγα καταστροφές. Θα ήταν λοιπόν καλό <clears throat> να η Επιτροπή να υποβάλει σε τεστ αντοχής τις παλιές υποδομές των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων. Κύριε Πρόεδρε, επ' αυτής της παραγράφου προτίθεμαι να προσθέσω κάτι ακόμα. Αν όλοι θεωρήσουμε ότι το έδαφος, η γη είναι η βάση. Άρα λοιπόν έχουμε μία φυσική υποδομή. Ε, προτίθεμαι να υποβάλω την ε, τροπολογία ότι σε φυσικές υποδομές όπου το έδαφος έχει υψηλή σεισμικότητα θα πρέπει να απαγορεύεται η οικοδόμηση, η οικοδόμηση πυρηνικών μονάδων. Είναι μέσα στις υποδομές και θεωρώ ότι το φυσικό περιβάλλον είναι υποδομές και θα πρέπει τουλάχιστον να δούμε ότι αποφεύγουμε ε, τον κίνδυνο μιας πυρηνικής καταστροφής σε σεισμογενή ε, περιοχή. Ευχαριστώ. Először Καταρχήν να πω πως ο εισηγητής ε, έκανε μια εξαίρετη εργασία και να τον συγχαρώ. Αλλά πρέπει να ομολογήσω πως μετά από το ατύχημα της Φοκοσίμα τα επίπεδα ασφάλειας έχουν ε, αυξηθεί. Ορισμένα κράτη-μέλη συναγωνίζονται σε θέματα πυρηνικής ενέργειας. Ως εκ θα πρέπει να ενισχύσουμε και να εξυγχρονίσουμε τις ενεργειακές υποδομές, να μειώσουμε στο ελάχιστο την εξωτερική μας εξάρτηση. Θα πρέπει θα αναφερθώ στο ευάλωτο της Ανατολικής Ευρώπης για τον ενοφοδιασμό στις ε, αέριο. Πρέπει απαραίτητα να καταγράψουμε πρόοδο σημαντική, να δημιουργήσουμε δίκτυα που θα λειτουργούν αποτελεσματικά, ιδιαίτερα σε όλη φορά τι διασυνδέσεις σε διασυνοριακό επίπεδο και να προωθήσουμε την, την ενεργειακή απόδοση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από ορισμένους ε, ενεργειακούς φορείς αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να επικεντρωθούμε και στις δικές μας ε, δυνατότητες και πόρους. Ε, Κανένα μου, οι υποδομές ε, αερίου δεν αναφέρονται εκτενώς στην έκθεση, γι' αυτό και εγώ καταθέτω τροπολογίες. Πρέπει να επικεντρώσουμε επίσης την περιφερειακή συνεργασία, προκειμένου να εγγυηθούμε τον ανεφοδιασμό σε αέριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο σκιώδης εισηγητής ο κύριος Ζαντό ε, δυστυχώς ε, αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι σε μια συζήτηση των συντονιστών της ΙΝΤΑ. Μου ζήτησε όμως να ευχαριστήσω τον κύριο Σόζα για τη συνεργασία και να σας μεταφέρω κάποια σχόλια. Τρία σημεία θα ήθελα να αναφέρω σύντομα. Πρώτα απ' όλα έχουμε σοβαρές αμφιβολίες κύριε Σόζα Βάγνερ για το εάν κάποια άλλη μορφή φυσικού αερίου ή δέσμευση άνθρακα ε, έχουν κάποιο νόημα όταν μιλάμε για το 2020. Ίσως παραπέρα, αλλά δεν θεωρούμε εντός αυτού του χρονικού ορίζοντα δεύτερον. Καλό θα ήταν και ξέρω πώς εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση να μην κάνουμε το λάθος σε αυτή την έκθεση που είχαμε κάνει στα 10E. Να κάνουμε δηλαδή έναν μεγάλο κατάλογο διαφόρων κριτηρίων και στο τέλος να μην βγει τίποτα. Πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι. Τρίτον, και κάνατε μία πρόταση που είναι πάρα πολύ καλή, την πρόταση μιας ιεραρχίας υποδομών, δηλαδή σαφές προτεραιότητες. Να προσπαθήσουμε πρώτα απ' όλα να δούμε είναι κάτι αναγκαίο, μετά να προσπαθήσουμε να ανακαινήσουμε κάτι και μετά να έχουμε νέες κατασκευές. Πράγματι, ε, συμφωνούμε πάρα πολύ με αυτό και σας ευχαριστούμε άρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Καρβάλια. Thank you, Chair. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι συνάδελφοι έκαναν πολλές παρατηρήσεις με τις οποίες συμφωνώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή μας, τον κ. Σοζαβάνη θα ήθελα να σχολιάσω δύο ζητήματα που σχετίζονται με τροπολογίες που συνυπέγραψα με κάποιους συναδέλφους. Πρώτον, η σημασία ε, της χρήσης ε, της υποδομής ε, που υπάρχει στην εμπειρική Χερσόνησο και για τροφοδότηση των Πυρηναίων. Ε, υπάρχουν 7 μονάδες στην Ιβηρική Χερσόνησο και η ενίσχυση των διασυνδέσεων με τα λοιπά δίκτυα της ε, Χερσονήσου θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εφοδιασμό ε, της κεντρικής ε, νοτιού και ανατολικής Ευρώπης. Τέλος, εγώ προτείνω μια τροπολογία βάσει της οποίας τονίζεται η ιδιαιτερότητα ε, των ενεργειακών υποδομών των απομονωμένων νήσων. Χιλιάδες νησιά υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 9 εξόχως απόμακρες, ε, ε, εξόχως περιοχές που έχουν ενεργειακές υποδομές στις οποίες θα πρέπει να διασυνδέσουμε τα υπόλοιπα δίκτυα. Έχω υποβάλει μαζί με άλλους συναδέλφους διάφορες τροπολογίες που σχετίζονται με αυτά τα ζητήματα και ελπίζω να συμφωνήσουν και να με υποστηρίξουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Η κυρία Φιγκυρέιντο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, και εγώ θεωρώ πως ε, ε, το ότι έχουν κατατεθεί τόσο πολλοί άριθμες τροπολογίες καταδεικνύει το ενδιαφέρον όλων των χωρών για αυτό το ζήτημα. Συζητούμε τώρα ε, το θέμα των ενεργειακών υποδομών που έχουν κέρια σημασία για την οικονομική ανάπτυξη. ενέργεια έχει καταλητικό ρόλο για την οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Και γι' αυτό έχω υποβάλει τροπολογίες με τις οποίες προσπαθώ να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτά τα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας ε, και ε, για την ανάγκη ε, αυξημένου δημοσίου ελέγχου αυτού του τόσο σημαντικού τομέα. Πρόκειται για πολύ σημαντικές επενδύσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα θα πρέπει να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες μας στον ενεργειακό τομέα, τους ώστε ο ανεφοδιασμός να εξασφαλιστεί με την μικρότερη δυνατή εξάρτηση για να κατοχυρώσουμε αυτήν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Ε, μάθαμε από την Ιαπωνία ότι χρειάζεται αυξημένους δημόσιος έλεγχος. Ε, σε όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να αυξηθεί ο έλεγχος ή τουλάχιστον στα κράτη-μέλη όπου υπάρχουν τα σοβαρότερα προβλήματα. Και κάποιε από τις τροπολογίε που υπέβαλα σχετίζονται με αυτές τις ανησυχίε που μόλις εξέθεσα. Συμφωνώ με αυτά που είπε η συνάδελφο σχετικά με την κατασκευή των πυρηνικών ε, μονάδων. Θα πρέπει να αποφύγουμε τους ε, σοβαρούς κινδύνους, την ε, οικοδόμηση τέτοιων μονάδων σε περιοχές κινδύνου, αντλώντας διδάγματα από τις πολύ αρνητικές εμπειρίες που είχαμε, όπως αυτή της Ιαπωνίας, αλλά δεν είναι και η μοναδική. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα δύο ζητήματα, δηλαδή η οικοδόμηση νέων πυρηνικών μονάδων θα πρέπει να λαμβάνει τον κίνδυνο που διατρέχουμε σε διάφορα επίπεδα, αλλά και το θέμα του ελέγχου δεν θα πρέπει να συσχετίζεται μόνο με το κέρδος, θα πρέπει να κατοχυρώσουμε ένα δημόσιο έλεγχο, ούτω ώστε να μην διατρέξουμε ε, αυτό το σοβαρό ε, κίνδυνο του πυρηνικού ατυχήματο, γιατί τον κίνδυνο τον διατρέχουν όχι μόνο άνθρωποι, αλλά ολόκληρες ε, περιοχές, ολόκληρες χώρες, ολόκληρα τμήματα υπήρου μπορούν να πληγούν από ένα τέτοιο ατύχημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα σύντομα η Κομισιόν, αλλά σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας είπα βεβαίως. Ε, εντάξει. Ε, είμαι ακόμα εντυπωσιασμένο από την παρουσία του κυρίου Επιτρόπου. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Σόζα Βάγνερ για την εκθεσή του. Είμαστε ικανοποιημένοι. Συνεχίζεται ούτω ή άλλω ο διάλογό μα και νομίζω ότι είναι υποφελή για όλου. Τέσσερι μόνο παρατηρήσει θα κάνω, Πρόεδρε. Πρώτον, Ελπίζω ότι ο κύριος Σόζα Βάγκνερ θα μπορούσε να τροποποιήσει κατά τη τροπολογίες σχετικά με τις προτεραιότητες, όπως και ο κύριος Κόφερ, ανησυχώ κι εγώ, διότι νομίζω ότι είχαμε ε, συμφωνήσει για τους μεγάλους ε, διαδρόμους Ελπίζω λοιπόν να είναι καλή η συμβολή του Κοινοβουλίου για τα κριτήρια επιλογής μεμονωμένων προγραμμάτων. Δηλαδή, ε, ενσωμάτωση στην αγορά, ασφάλεια ανεφοδιασμού, τέτοια πρέπει να είναι τα κριτήρια μας. Ή όπως είπε ο κύριος ε, Κάρες, ε, εξάρτηση από μία μόνο πηγή, ενεργειακή απόδοση των νεώσιμων πηγών ενέργειας, στόχοι για τη μείωση των εκπομπών κτλ. Αυτά τα κριτήρια είναι σωστά, αλλά πρέπει να αποφύγετε και παρόλα όλα αυτά έχουν ήδη κατατεθεί τέτοιε τροπολογίε. Πρέπει να αποφεύγονται λοιπόν όταν αφορούν σε ένα μόνο πρόγραμμα, διότι θα πέσουμε στην ίδια παγίδα. Όπω όταν συζητούσαμε τελευταία φορά αυτό το ζήτημα, είχαμε ε, ένα τεράστιο αριθμό προγραμμάτων χωρί καμία προτεραιότητα. Οπότε εστιάστε παρακαλώ την προσοχή σα στα κριτήρια επιλογή των μεμονωμένων προγραμμάτων. Δεύτερον, ε, είμαστε ευγνώμονες διότι ο συγητής ε, τόνισε τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας ε, ως προς την επιλογή των προγραμμάτων. Έχουμε θετικές εμπειρίες για τη Βαλτική θάλασσα, παραδείγμα του χάρη για τις χώρες ε, της ε, Βόρειου θάλασσας. Είναι ομάδα ε, υψηλού επίπεδου για τις ενότιες διασυνδέσεις δικτύων και νομίζω ότι είναι στο σωστό επίπεδο αυτή η ομάδα για να συζητάει, να εξετάζει αυτά τα προγράμματα. Οπότε όλες οι σχετικές τροπολογίες προς επίρρωση δηλαδή της συνεργασίας είναι ευπρόσδεκτες. Τρίτον, δεν θέλουμε να είμαστε επικριτικοί για τη συνενετική λύση σχετικά με την αδειοδότηση τη... Με ζητούν κάποιοι καλύτερη εναρμόνιση, χρειάζονται νέε διαδικασίε, μα είπαν. Συμφωνούμε. Επίση, τα ενιαία σημεία επαφή, αυτέ οι μονοαπευθυντικέ θηρίδε, ε, νομίζω είναι ιδέε που ευθυγραμμίζονται με την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλο, ε, ρύθμιση τη αγορά και χρηματοδότηση. Ε, πολύ υποστηρίζεται τις ιδέες μας ε, και υποστηρίζεται και τα μέσα που ε, δημιουργήσαμε μέσα από τις διάφορες νομικές πράξεις για την ενιαία αγορά, για τα τέλη, την ετοιμολόγηση κτλ. Ε, κοιτάξτε, οι υποδομές ως επιτοπλίστων θα χρηματοδοτηθούν μέσα από τα εφιστάμενα μέσα, αλλά υπάρχουν και στην αγορά κάποιες ατέλειες και θα θέλαμε να τις ε, διορθώσουμε. Ε, Αυτά τα ομόλογα είναι ένα καλό ε, μέσο, αλλά θα πρέπει να φροντίσετε ώστε ε, να μην υπάρχει χρηματοδότηση των προγραμμάτων αλλά των εταιρείων. Δεν είναι πάντοτε η καλύτερη λύση η χρηματοδότηση των έργων για να χρηματοδοτήσετε τι δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Το corporate financing ε, μου φαίνεται καλύτερη λύση. Δηλαδή δεν χρειάζεται χρηματοδότηση μέσω ομολόγων όταν ζητάει μια εταιρεία κάποια επιδότηση και στο EPR φάνηκε ξεκάθαρα ότι μπορεί να είναι ένα καλό κίνητρο η χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δράσης. Ας αφήσουμε αυτό το ζήτημα και ας δώσουμε ρευστότητα στις επιχειρήσεις αντί να χρηματοδοτούμε μέσω συγκεκριμένων έργων ούτω ή άλλω η άλλω η χρηματοδοτηση θα πρέπει να προσαρμόζεται κατά περίπτωση στι ανάγκε ή του προγράμματο ή του φορέα τη επιχείρηση που έχει αναλάβει την εκμετάλλευση. Ευχαριστώ και τώρα θα ακούσουμε και πάλι τον εισηγητή. Να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στην συζήτηση για τα καλά τους λόγια, για τις υποδείξεις τους, να ευχαριστήσω και την Κομισιόν. Ξεκίνησα αναφερόμενο στην Θεία Κομμωδία και στην Θεία Κομμωδία αναφέρεται ότι στον, ε, στην κόλαση χάνει κανείς ε, την ελπίδα αλλά εγώ εδώ απέκτησα την ελπίδα ότι με τη βοήθεια των συναδέλφων θα, ε, θα πετύχω ένα καλό αποτέλεσμα. 26 Μαΐου θα ψηφίσουμε. Τελειώσαμε αυτό το θέμα. Περνάμε στο υπαριθμό 19. δηλαδή το νόμο περί μικρών επιχειρήσεων, κοινή δήλωση, θέλει κάποιος το λόγο, ο κύριος Μπέντσεν πρώτος, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίζω την αναθεώρηση του σχετικού νομοθετήματος από την Κομισιόν. Περιέχει αρκετές καλές ιδέες για το πώς θα βελτιωθεί η νομοθεσία και θα γίνει καλύτερη για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην κρίση μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αντιμετωπίζουν ακόμα σήμερα. Μέχρι στιγμή είχαμε επικοδομητικό διάλογο με όλα τα κόμματα εντός του Κοινοβουλίου. Έχουμε κάνει λοιπόν μια καλή αρχή για τις περαιτέρω συζητήσεις. Στο Στρασβούργο, το ΕΛΚ, το κομμάτι μας δηλαδή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συναντηθήκαμε με τον απεσταλμένο της Κομισιόν για τη, από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και νομίζω πως είχα μια καλή συζήτηση Με βάση αυτά λοιπόν έχω κάποιες ε, περαιτέρω παρατηρήσεις για το ψήφισμά μας. Είναι και η ώρα να αναλάβουμε δράση. Φτάνουν τα λόγια πρέπει να γίνουμε συγκεκριμένοι στο πώς θα βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καλωσορίζω τα τρία βασικά ζητήματα που ανέφερε η Κομισιόν. Δηλαδή μείωση της γραφειοκρατίας, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και πρόσβαση στις αγορές. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα για την απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υποστηρίζω βεβαίως την αρχή μία φορά να γίνονται τα πράγματα. Δεν πρέπει οι επιχειρήσει ε, να δίνουν τις ίδιες πληροφορίες σε διαφορετικές αρχές παραπάνω από μία φορά. Η ΔΕ Κομισιόν θα πρέπει να προωθήσει τη μείωση του διοικητικού άχθους γιατί ξέρετε πως δεν έχουν θέσει όλα τα κράτη-μέλη στόχους για τη μείωση. Χρειαζόμαστε πολιτική στήριξη. και χρειάζονται επιχορηγήσεις, εγγυήσεις και επιχειρηματικό κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει επίσης να δούμε πώς θα βελτιώσουμε την πρόσβασή τους στις δημόσιες προμήθειες. Πρέπει να βελτιωθεί ο διάλογος με τις ε, αρχές για να καθοδηγήσουμε τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμμετοχή τους στις δημόσιες προμήθειες. Πρέπει να δούμε το κατόφλι επίσης για τις ε, προμήθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αυξηθεί αυτό το κατόφλι τότε, εάν δηλαδή δεν υπόκεινται αυτά τα συμβόλαια στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορέσουν να κάνουν ευκολότερα προσφορές οι μικρομεσαίες αυτές οι επιχειρήσεις με λιγότερη γραφειοκρατία. Επίσης θα πρέπει να δούμε το πώς συμβάσεις θα δημοσιεύονται ε, προκηρύξεις, δηλαδή για να ε, γνωρίζουν ε, τις προσφορές που μπορούν να υποβάλουν οι επιχειρήσεις. Επίσης πρέπει να μειωθεί βεβαίως το διοικητικό βάρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην περίπτωση που κάνουν διασυνοριακές προσφορές. Οπότε ανησυχώ βεβαίως λίγο Ε, όταν μιλάμε για τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 99,8% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη καλύπτονται από τον υπάρχοντα ορισμό. Το να αναθεωρήσουμε τον ορισμό θα νερώσει το τι εννοούμε με τη λέξη μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νομίζω είναι αντίθετο με το πνεύμα του νομοθετήματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Να δώσω τον λόγο στην κυρία Χέρτσοκ. Α, όχι, έφυγε. Κυρία Χέρτσοκ, σας ενδιαφέρει να λάβετε το λόγο. Yeah, uh, in this debate, I think. Σας ενδιαφέρει η συζήτηση εκεί που είχατε. Όχι, όχι, γενικά με ενδιαφέρει. Όχι μόνο σήμερα. Πήγα να κάνω μια μικρή διαβούλευση. Με ξέρουν όλοι ότι ασχολούμαι με το Small Business Act. Δεν χρειάζεται να συστηθώ τώρα. I think it's a very, very important uh, that uh, the Commission. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εξέδωσε τώρα νέα πρόταση γιατί το κοινοβούλιο ε, στην τωρινή θητεία του έτσι, δεν είχε ακόμη την ευκαιρία να αποφανθεί για το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ήρθε η ώρα να κινηθούμε πριν εγκριθεί το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να να χρησιμοποιήσουμε και άλλα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω είναι σημαντικό να το πούμε. Ο κύριος Σταγιάννη και το επιτελείο του, λοιπόν, πολύ καλά έπραξαν και υπέβαλαν νέα πρόταση. Και πριν από έξι εβδομάδες, πριν από δύο μήνες, συναντήθηκε με τον εκπρόσωπο για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, δείτε τι επιτυχημένες ε, ιστορίες ε, του περσινού έτους, σίγουρα, ε, του, της περασμένης του Κοινοβουλίου. Σίγουρα το Small Business Act είναι μία από τις επιτυχίες και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συνεχίσει αυτή η ενάρετη πορεία και στο μέλλον. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι το πολιτικό μας έμβλημα μεταξύ άλλων αυτό το θέμα. 116 μέλη έχουν, ε, βουλευτές του Κοινοβουλίου έχουν υπογράψει ένα σχετικό έγγραφο που ο στόχο έχει να προαγάγει τη δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει να εργαστούμε, πρέπει να προχωρήσουμε. Κάτι άλλο εξίσου σημαντικό. Κάθε πολιτική σχετίζεται με την ε, στρατηγική 2020 Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα περιμένουμε και θα ξυπνήσουμε το 2019 και θα πούμε ουπ, σχεδόν εξέπνευσε η προθεσμία και δεν προλαβαίνουμε. Όχι. Χωρίς τα 23 εκατομμύρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων και χωρίς ε, τα 2 τρίτα ε, του εργατικού δυναμικού που εργάζονται σε ΜΜΕ δεν πρόκειται να τα καταφέρουμε, να υλοποιήσουμε καμία στρατηγική. Οπότε μέσω των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους θα συνεργαστούμε όλοι για να υλοποιήσουμε τους στόχους στρατηγικής 2020 γιατί πέντε από αυτούς τους στόχους έχουν ιδιαίτερη σημασία και θα ήθελα να ενταχθούν ε, στο νέο έγγραφο για το Small Business Act. Πώς, με ποιο τρόπο, τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να μοιράσουμε ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα την ενεργασία που πρέπει να κάνουμε για τα, την έρευνα και τα ερευνητικά πρόγραμματα. Είπαμε σήμερα το πρωί τι κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε για τι τις κλιματικές αλλαγές, για την παιδεία, για την καταπολέμηση της φτώχεια και για την ε, πρόθεση τη απασχόληση. Και τέλος τι μπορούμε να κάνουμε για τις ε, ανθούσες ε, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λοιπόν, η ενιαία αγορά έχει τεράστιο δυναμικό, το οποίο δεν έχουμε αξιοποιήσει ακόμη πλήρως και άρα θα πρέπει να ε, αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας προσφέρει η ενιαία αγορά, κυρίως ως προς τις ΜΜΕ. Ο κόσμος των ΜΜΕ, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πλήγεται πλήττεται από την αγορά κρατικών προμηθειών, διότι δεν υπάρχει πάντοτε ισότιμη μεταχείριση ανάμεσα στι μεγάλε επιχειρήσει και τι μικρομεσαίε. Πάντω, ναι, οι κρατικέ προμήθειε είναι σημαντική αγορά, οπότε θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στι κυβερνήσει των κρατών μελών και στις ε, αυτοδιοικητικές αρχές ε, ε, για να συμπεριλάβουν στο παιχνίδι αυτό του ανταγωνισμού και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ε, βέβαια θα σας πούν ότι δεν έχουν πρόσβαση, ε, έχουν μόνο περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα θα πρέπει να συνεχίσουμε να δρούμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ξέρετε, πέρα από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση υπάρχει και η πρόσβαση στις γνώσεις. Οπότε το μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι αυτό ακριβώς. Να αναγνωρίσουμε το δικαίωμα καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ε, να εφαρμόζουμε την καινοτομία μέσω των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα αναφέρουμε στο Small Business Act. Επίσης, τις αδυναμίες μας ε, πρέπει να τις σχολιάσουμε, να τις αναφέρουμε. Υπάρχει ακόμη διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλλα και οφείλουμε να κάνουμε κάθε τι περνάει από το χέρι μας για να συμμετάσχουν ισότιμα και οι γυναίκες και οι άντρες. Δεν υπάρχει κανένας αντικειμενικός λόγος που να αιτιολογεί τη μη συμμετοχή των γυναικών, άρα θα πρέπει να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο και υποστηρίζουμε και παρακινούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε όλες τις προσπάθειες που κάνει για να ε, ενισχύσει ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι ποτέ δεν θα συμφωνήσουμε με την ε, περικοπή των ε, δαπανών, των ανθρωπίνων πόρων, ε, των θεσμικών δυνατοτήτων προσφέρονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτός είναι ο αγώνας μας και είτε μιλάμε για έρευνα, για καινοτομία, είτε για οτιδήποτε άλλο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την πάγια θέση ότι θέλει να προστατεύσει τον κόσμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να αυξήσει το ρόλο τους γιατί έχει καταδειχθεί η σημασία τους. Εάν τα ξεχάσουμε όλα αυτά, θα έρθουμε αντιμέτωποι με τον ευρωσκεπτικισμό. Ας μην κρυβόμαστε, διότι αν αφαιρέσουμε αυτά τα μέσα που είναι διαθέσιμα τώρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα διωγγωθεί ο ευρωσκεπτικισμό. Δεν είναι η σωστή στιγμή να κάνουμε τώρα περικοπές, το αντίθετο πρέπει να κάνουμε να επιταχύνουμε πρέπει σε σχέση με το παρελθόν, ούτω ώστε να συμμετάσχουν ισότιμα οι μικρομεσαίε επιχειρήσει στην ενιαία αγορά και να έχουμε και άλλες τέτοιες επιτυχημένες ε, ε, ιστορίε ε, στην Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρώ πως πρόκειται για μια πρωτοβουλία ιδιαίτερα σημαντική Αυτά που είπε ο κύριος Μπέντσεν ε, είναι πολύ σημαντικά. Εδώ και χρόνια υπάρχουν τεράστιες δυσκολίε και ιδιαίτερο ε, διοικητικό άχθος ε, για την διαχείριση επιχειρήσεων. Φυσικά αυτό εξαρτάται από χώρα σε χώρα και η μόνο ευθεντική θηρίδα αναφίβολα βοηθάει τόσο τις μεγάλες όσο και τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε διάφορες ε, συζητήσεις που είχαμε εξετάσαμε τις δυνατότητες που υπάρχουν για να ξεπεράσουμε την ε, κατάσταση και τα προβλήματα και παρατηρούμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες δυσκολίες προκειμένου να προσφεύγουν σε, σε, δανεισμό και στην ε, χρηματοδότηση μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ε, επί του εξής σημείου. Εάν δεν ε, λειτουργούν ε, μικρές περιφερειακές τράπεζες, οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες ε, δεν θεωρούν ότι είναι σημαντικοί συνομιλητές και πελάτες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να περιπλέκει περαιτέρω τα πράγματα και να δυσκολεύει την ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ας αφήσουμε τις ε, προθεσμίες οι οποίες είναι πολύ μεγάλες ως ε, βουλευτές. Χρειάζεται να στείλουμε ένα μήνυμα προς τις ε, επιχειρήσεις αυτές και να τονίσουμε πως εδώ πρόκειται για ένα στοιχείο αθέμητου ανταγωνισμού που πλήττει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τώρα. Αναφορικά με τις επιμέρους υπηρεσίες, εμείς ζητάμε να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των ε, μικροψηφίων επιχειρήσεων και των ε, πιστοτικών ιδρυμάτων προκειμένου να έχουν μια καλύτερη πρόβαση στην ε, χρηματοδότηση διότι βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά αντιμετώπιση μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων από τα τραπεζικά ιδρύματα. Οι αλλαγές οι οποίες έγιναν σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης ε, αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, π.χ. οι εγγυήσεις οι οποίες θα πρέπει να παρέχουν έχει ως αποτέλεσμα πολλές αυτές τις επιχειρήσεις ε, να μην μπορούν να προσφεύγουν σε αυτές τις ε, αγορές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο συνεχίζει να εφίσταται. Δεν πρέπει να υπάρχουν οι ίδιες απαιτήσεις και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά τα σχέδια χρηματοδότησης ε, χρειάζεται να αναλυθούν ε, περαιτέρω, διότι αναφίβολα είναι δραστηριότητες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, ειδικά όταν αυτές διεξάγονται με την απαραίτητη διαφάνεια αλλά στην περίπτωση αυτή μιλάμε για θέματα ανταγωνισμού που προκύπτουν μεταξύ των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων και φυσικά αυτές οι οποίες ε, επηρεάζονται αρνητικά είναι οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στα πλαίσια λοιπόν της ε, διαδικασίας ε, σύστασης ε, νέων επιχειρήσεων θα πρέπει να φροντίσουμε να χορηγείται μια ιδιαίτερη προσοχή και βοήθεια σε αυτές τις επιχειρήσει. επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ και εγώ και να κάνω και εγώ μια παρατήρηση όσον αφορά την σημασία της, ε, με το επιχειρήσεων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, όπου συμφωνούμε ότι δεν είναι ικανοποιητικά. Αλλά αυτό το οποίο με ενοχλεί και πρέπει να μας απασχολήσει και στην Κομισιόν τι θα κάνουμε συγκεκριμένα. Γιατί να λέμε πόσο σημαντικό είναι και πρέπει να κάνουμε περισσότερα δεν χρειάζεται. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα. Αλλιώς δεν θα βοηθήσουμε κανέναν. Σας ευχαριστώ να υπενθυμίσω πως μέσα Μαΐου θα έχουμε στην Ολομέλεια και το ψήφισμα και την προφορική ερώτηση και έτσι να δώσουμε μια πολιτική όθηση στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελείωσε αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Τελείωσε άρα η ημερήσια διάταξη για σήμερα και τα λέμε αύριο το πρωί. Γεια σας.